Καλημέρα σας. Δεν νομίζω να έχουν έρθει όλοι εγκαίρως για το πρώτο θέμα, αλλά είμαστε αρκετοί ήδη. Και έχουμε ένα σχέδιο μερικής διάταξης, με αυτό θα ξεκινήσω. Μία η αλλαγή που αφορά την ψηφοφορία για την έκθεση Γκοζές ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθεται σε κυκλοφορία δεν θα ψηφιστεί διότι η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων ακόμη δεν έχει καταθέσει την γνωμοδότησή τη. Και άρα πρέπει να περιμένουμε. Θα ψηφίσουμε σε κανένα δύο εβδομάδες ακόμα. Δεν νομίζω να έχει κανεί αντίρρηση. Είναι ούτω ή άλλως καλύτερο να περιμένουμε τη γνωμοδότηση επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Θα έχουμε λίγο χρόνο. Περιθώριο αργότερα στην ε, διάρκεια των ψηφοφοριών. Καταλαβαίνετε ότι ο ενδεικτικό, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχουμε δεν θα τηρηθεί. Θα είμαστε έτοιμοι νωρίτερα γιατί, για να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Και έτσι προχωρώ στο σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Επινγκ. στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. ΔΕΡΚ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφέτο τον Ιούνιο η Επιτροπή υιοθέτησε την πρότασή τη, ε, την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη δικασία μακροοικονομικών ισορροπιών. Θα ήταν σκόπιμο βεβαίω να έχουμε πρώτα ε, νομοθεσία για την ποιότητα των στατιστικών και μετά το MIP τις μακροοικονομικές ανισορροπίες δηλαδή, αλλά όπως παραδοσιακά γίνεται, ξεκινάμε από κάτω και μετά πάμε προς τα πάνω. Και έτσι θα εξετάσω την πρόταση της Επιτροπής με μια καρτεσιανή, αυστηρά καρτεσιανή προσέγγιση, όπως λέμε και στα γαλλικά. Και έτσι κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στο γενικό στόχο του προτινόμενου κανονισμού, την ενίσχυση λέει, δηλαδή, της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και βέβαια χρειαζόμαστε γι' αυτό ένα ε, βελτιωμένο σύστημα ε, παρεκολούθησης της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, δι, δέλτα Χρειάζεται να αναπτυχθούν σαφεί απαιτήσει και διαδικασίε, να είμαστε προσαρμοσμένοι καλύτερα στις ισχύουσε διαδικασίε των στατιστικών και να ευθυγραμμιστεί ώστε να καλυφθεί και το κομμάτι που λείπει από το μοσαϊκό αυτό. Γι' αυτό θέλω να προχωρήσω στο δυνατόν παράλληλα με το πλαίσιο της ΔΕΛΤΑ Προτείνω ως εκ τούτου πρώτον τον περιορισμό της ε, επιβολής κυρώσεων μόνο στις χώρες του ευρώ, όπως συμβαίνει και στο πλαίσιο της ΔΜΑ. Δεύτερον, οι αδίποτε πρόστιμα συλλέγονται θα πρέπει να ε, αποδίδονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και όχι στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ακριβώς όπως συμβαίνει και στη ΔΜΑ. Τρίτον, νομική βάση βλέπω ότι το άρθρο 338 μπορεί να ε, παρουσιάζει νομικά προβλήματα ως νομική βάση για τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Και γι' αυτό έχω συμπεριλάβει και ένα, μια αιτιολογική σκέψη όπου ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει με μια πρόσθετη νομική βάση εφόσον χρειαστεί επί παραδείγματι το άρθρο 121 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την οικονομική διακυβέρνηση πάνω στην οποία επίση μεταξύ άλλων ε, βασίζεται και η ΑΛΦΑ Και επίσης αναφέρομαι σε μια ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τις πρακτικές για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Δεν σκοπεύω να επανειφεύρω τον ε, τροχό. Αξιοποιώ λοιπόν ε, κείμενο από την έκθεση του συναδέλφου Walk για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Επί παραδείγματι, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα ΕΣΣ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ΕΣΣΚΤΑΦ είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση στατιστικών με στοιχεία που ε, αφορούν τη ΔΜΑ. Σε αυτά στηρίζεται δηλαδή η ΔΜΑ και όπως αναφέρει και ο συνάδελφος Γουόγκ, είναι απαραίτητο να υπάρχει και στενή συνεργασία μεταξύ των δύο συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή Στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, ΕΣΝΙΧΙ θα μπορούσε να προσφέρει, λόγω τη εμπειρία τη στον τομέα των στατιστικών, συμβουλές όσον αφορά τις πρακτικές λειτουργικές ρυθμίσεις για μια τέτοια συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων. Επίσης, το, η ΔΜΑ έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία Τη ΕΚΤ και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάγεται στις ίδιες ε, προϋποθέσεις ε, και πρακτικές διαφάνειας και λογοδοσίας με κάθε άλλο όργανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης πιστεύω ότι ο οικονομισμός θα πρέπει να προσδιορίσει την επακριβή διαδικασία μετάδοσης των δεδομένων και συγκεκριμένα προτείνω να οριστεί μια δίλη ημέρα την οποία, κατά την οποία θα αποδίδονται τα στοιχεία, θα βγαίνουν δηλαδή από την Eurostat και έτσι θα ε, ικανοποιείται ο, ο στόχος της ε, καταγραφής, ταυτόχρονης καταγραφής. Δεύτερον θα υπάρχει μια δίλη ημέρα δημοσιοποίησης, ώστε να ενημερώνεται και ο υπόλοιπος κόσμος για να εξυπηρετηθεί ο στόχος της ασφάλειας για τις λεγόμενες αποστολές και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Βλέπω πεδίο για βελτίωση. Και έτσι προτείνω συγκεκριμένα να ανα επανονομαστούν αυτές οι αποστολές σε επισκέψεις διαλόγου Επίσης, και μια και είμαι και διαμαρτυρόμενο. Η λέξη αποστολή θα πρέπει να σας πω, μου θυμίζει οι αραποστολές, οι ε, ε, προσελητισμού από το Βατικανό. Ή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κιόλας την ιδέα τη της αποστολή. Λοιπόν, αυτές οι αποστολέ δεν έχουν να κάνουν ούτε με εισβολή, ούτε με προσελητισμό, αλλά με μια ε, αξιολόγηση από του ομολόγου και διάλογο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέψεις διαλόγου. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ επισκέψεων διαλόγου και οδήποτε άλλων ερευνών που μπορεί να οδηγούν σε άλλα αποτελέσματα. Επίσης προτείνω να εμπλέκεται έγκαιρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκ του σύνεγγε στη διαδικασία αυτή. Ιδιαίτερα η δική μα Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί σε συζήτηση και ακροάσει στου επικεφαλεί των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Προσβλέπω δε στην επικοδομητική συνεργασία στο θέμα αυτό με του συναδέλφου, την ελπίδα να καταλήξουμε σε μια καλή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους πιο εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριο Ντόρφμαν. Thank you, Ja, äh, ich denke, ähm, ich kann mit vielen... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τα περισσότερα που όσα είπε ο συνάδελφό. Η... Εξασφάλιση καλών στατιστικών είναι βέβαια προϋπόθεση και για την μακροοικονομική εποπτεία. Δεν συμφωνώ 100% στην ιδέα ότι πρώτα ξεκινάμε και χτίζουμε τη στέγη και μετά τα θεμέλια, επειδή θέλουμε να αναφερθούμε στις μακροοικονομικές προοπτικές. Νομίζω ότι οι καλές στατιστικές, τα καλά στατιστικά δεδομένα είναι μια πολύ καλή βάση και προϋπόθεση για να λειτουργήσει η μακροοικονομική εποπτεία. Και στο πλαίσιο άλλωστε του six packs της, της δέσμης εξημέντρων έχουμε ήδη εισαγάγει την ιδέα αυτή της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο κανονισμός, ο νέος αυτός κανονισμός, είναι απαραίτητος, είναι σκόπιμο να εισαχθεί. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία που έθιξε και ο κύριος Έπινγκ. Ε, παραδείγματι το θέμα του πιο επακριβούς ορισμού των επισκέψεων και ελέγχων στις αστικές υπηρεσίες ε, είναι απαραίτητο να προχωρήσει. Ε, η υποχρέωση για τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να διαθέτουν εγκαίρως στοιχεία είναι επίσης πολύ σημαντική και πρέπει να βελτιωθεί. Συμφωνώ να συνδυαστεί αυτός ο κανονισμός με τον σχετικό με το six ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος της διευκρίνησης του ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία, για να γνωρίζουμε δηλαδή στο ΣΥΚΣΠΑΚ μετά όλες τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις μεγάλες ε, συζητήσεις για τον ορισμό του τι είναι απαραίτητο στοιχείο ή κριτήριο για την επεξεργασία και για την μακροοικονομική προοπτική ε, και μια έχουμε, και έχουμε κάνει όλη πρόοδο στο six θα πρέπει αντίστοιχα να παρακολουθήσουμε εν ώψη της μακροοικονομικής εποπτείας την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων. Δεν μπορώ όμως να συμφωνήσω με την ιδέα στον κανονισμό αυτό να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των κρατών του, της ζώνης του ευρώ και των κρατών που δεν ανήκουν σε αυτό στην Ευρωζώνη. Η ποιότητα των στατιστικών πρέπει να αφορά και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, δεν μπορούμε να έχουμε διπλέ ταχύτητε εδώ ή μεταχείριση διαφορετική για το κάθε κράτο μέλο. Σε τελευταία ανάλυση, εφόσον δεν προκύπτουν και κυρώσει για τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει λόγο να υποβιβάσουμε την ποιότητα, την απαιτούμενη ποιότητα για τι στατιστικές αυτέ. Ανεξαρτήτως του αν ανήκουν στην Ευρωζώνη ή μη τα κράτη αυτά. Είναι βέβαια σημαντικό στο θέμα των κυρώσεων πάλι να παρακολουθήσουμε το πνεύμα και το γράμμα του Sixpack με την ε, αντίστροφη ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία με ένα μοντέλο σε δύο βήματα. Παραδείγματι την προειδοποίηση ή όχληση και μετά την κύρωση αυτή καθεύτη. Και νομίζω το ποσό μπορεί να είναι 0,05% έως 0,05% επί του ΑΕΠ, ένα ποσοστό αντίστοιχο και με αυτό που ε, προκύπτει από το ΣΥΚΣΠΑΤ για την Κεντρική Τράπεζα συμφωνώ με τον εισηγητή όταν ε, πρόκειται για στατιστικά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από ε, ενστάσεις απορρίτου και εμπιστευτικότητα των στατιστικών στοιχείων. Δεν μπορεί δηλαδή να παραβλαπτεί από αυτό η διαφάνεια των στατιστικών μας στοιχείων. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι μια έκθεση, πιστεύω, η οποία μπορεί ωραιότατα να μας οδηγήσει σε ένα πολύ καλό κοινό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Χουαν Κόκ. Ε, ε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του για ένα θέμα που εκ πρώτης όψεως ε, φαίνεται ίσως και βαρετό, ανιαρό, αλλά δεν ε, ε, είναι άμερο πολιτικής σημασίας. Αρχικά δημιουργήσαμε το εξάπτυχο ε, και μετά το συντονισμό των ε, οικονομικών πολιτικών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα προβλέπονται κυρώσει σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που στηρίζονται σε στατιστικούς δείκτες. Οπότε αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Και η χορήγηση αυτών των δικτών των στατιστικών θα πρέπει να γίνεται με το πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη συγκεκριμένη νομοθεσία που στόχο έχει την αναθεώρηση του κανονισμού πλαίσιου τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, αυτή η αναθεώρηση είναι όμοιρος, έχει γίνει όμοιρος μιας προσπάθειας και διαμάχης που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιας σύνδεσης που γίνεται. Ε, και μάλιστα προτάθηκαν ε, κυρώσεις κατά των ε, χωρών που εσκεμμένα παραποιούν τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν είχαμε νομική βάση για την επιβολή τέτοιων κυρώσεων. Είχαμε όμως συμφωνήσει με την Προεδρία του Συμβουλίου ότι αυτό το σημείο θα το καλύπταμε στην συγκεκριμένη τομεακή νομοθεσία για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα προτείνει την επιβολή κυρώσεων, χωρί όμω την κατάλληλη νομική βάση. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή που αντιμετώπισε αυτή τη δυσκολία στο σχέδιο έκθεσή του, προτείνοντα μια εναλλακτική νομική βάση αντί να παραιτηθεί πλήρω από αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιβολή κυρώσεων. Συμφωνώ με το στόχο του και με την προσπάθειά του, αλλά διαρωτώ με ένα σκόπιμο να περιορίσουμε τι κυρώσει μόνο στα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη, μια και το 121 αναγνωρίζεται ω νομική βάση και το 121 αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε εκτό Ευρωζώνη. Τώρα, ο εισηγητής θέλει να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της ε, Eurostat. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και εμείς στεναρά αυτή την πρόταση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να υπογράψουμε πολλές επιταγές σε λευκό μέσω διατάξεων που προβλέπουν εκτελεστικές και καταξιοδότηση πράξεις. Δεν ξέρω ε, αν είναι σκόπιμο να δεχτούμε αυτή την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μάλλον ε, είμαι κατά, θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Αντίθετα, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αποστολές στις χώρες μέλη, εκεί που αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότητας, δεν έχω αντίρρηση. και ο εισηγητής προτείνει απλές επισκέψεις διαλόγου. Προτιμώ την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να εμβαθύνουμε στη συζήτηση για όλα αυτά τα σημεία και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουμε σε πολύ καλή συμβαστική λύση για την έκθεση σας, κύριε Έπιγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Υπάρχει άλλος και ο καταρχήν. Ναι, ο εκπρόσωπος των Πρασίνων. Σκιώδης ηγητής είναι ο Φίλιμ Πλάμπερς. Θα διαβάσω λοιπόν τα σχόλιά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή του προσπάθεια ε, είμαστε υπέρ ε, των περισσότερων προτάσεων της έκθεσης, όπως διερεύνηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ε, στις τροπολογίες 15 και 24 και η, με, η μετατροπή των επισκέψεων σε, σε αποστολές έρευνας. Επίσης, την τροπολογία 19 για την υποστήριξη των θέσεων και την αναδιατύπωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συστάσεις που προτείνει η τροπολογία 21 καθώς και τη νομική εξουσιοδότηση που ζητάει η τροπολογία 22. Με όλα αυτά συμφωνούμε. Έχουμε όμως σοβαρές αμφιβολίες ως προς την αναλογικότητα της αρχικής πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι ένα πιο σταδιακό σύστημα όπως αυτό που αναφέρεται στο εξάπτυχο πακέτο, που μιλάει για την περίοδο της διόρθωσης των αιτιών που οδηγούν σε ανακριβή και αναξιόπιστα στοιχεία και μετά την υποβολή προειδοποίησης στα κράτη-μέλη και της απέτησης υποβολής διορθωτικού σχεδίου. Επίσης, θα προτιμούσαμε τα έσοδα από τα πρόστιμα να περιέρχονται στο κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως αρχικά πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Δεν βλέπω να θέλει άλλος κανείς το λόγο. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου για την υποστήριξη ε, που εκφράσατε για την έκθεση του κυρίου Έπινγκ, ε, όπως προέκυψε από τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση και θεωρεί ότι ένα εύρωστο σύστημα ε, παρακολούθησης των στατιστικών ε, στοιχείων είναι απαραίτητο και για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και για το εξαπλό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά και τον εισηγητή και τα μέλη της ΕΚΟΝ για τις προσπάθειές σας. Θα ήθελα τώρα συντομία να αναφερθώ σε μερικά σημεία της έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι οι παραποίησεις των, ε, το στατιστικών στοιχείων είναι απαράδεκτες. Η σκόπιμη υποβολή ανακριβών στοιχείων θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουν τα κράτη-μέλη από την σκόπιμη υποβολή τέτοιων στοιχείων και αυτό το λόγο έχουν και οι κυρώσεις. Βέβαια μπορούν να γίνουν κάποιες παραποίησεις στατιστικών στοιχείων και εντός και εκτός ευρωζώνη. Ω εκ τούτου, στην πρότασή μα θεωρούμε ότι η πρόταση θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και να μην περιορίζεται μόνο στα μέλη της Ευρωζώνης. Η εφαρμογή των κυρώσεων σε όλα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην πρόταση τα έσοδα από τα πρόστιμα να περιέρχονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό, μια και θα ε, εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο θέμα αφορά τη νομική βάση. Σημειώσαμε προσεκτικά τα σχόλιά σας και σίγουρα θα συνεχίσουμε την εξέταση αυτού του τεχνικού, νομικοτεχνικού ζητήματος σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τις αποστολές ή τις επισκέψεις στα κράτη-μέλη. Στόχος μας είναι Αποκινούμε τα κράτη-μέλη να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Θέλουμε να αποφύγουμε επικαλύψεις και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας ε, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα, Στατιστικό Σύστημα και το, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών προκειμένου να ελοπίσουμε αυτό το στόχο. Η δυνατότητα όμως ε, διενέργειας αποστολών όπου δει και όπου δεν αρκεί το μερική νομοθεσία για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, τέτοιε αποστολέ θα μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα και προσβλέπω σε συνέχιση της στενής συνεργασίας με την ΕΚΟΝ προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων για τις στατιστικές πληροφορίες και αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Έπινγκ, τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Καταρχήν, ως προς την παρατηρήση του κυρίου Ντόρφμαν για την εφαρμογή του κανονισμού, ο κανονισμός για τη ποιότητα των στατιστικών ισχύει, για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν περιορίζεται δηλαδή στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μόνο. Τώρα, εγώ μίλησα εκ παραλλήλου για τη διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και αυτή η διαδικασία ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Εκεί έγκυται η διαφορά η εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών ε, καλύπτει ολόκληρη την Ευρωζώνη, οι κυρώσεις περιορίζονται μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό προβλέπει η ισχύουσα διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ευχαριστώ και τον κύριο Χουανκόγκ και τις παρατηρήσεις του. Έχουμε ξανασυζητήσει σε σφοδρέ ε, συζητήσει ε, το θέμα των στατιστικών, γιατί για μα είναι συναρπαστικά αυτά τα θέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ανησυχίε για τη νομική βάση, είναι εύλογε. Ε, και χαίρομαι που αναγνωρίζει το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει προθυμία για την αντιμετώπιση του. Ο κύριος ε, Γκίγκολτ ε, ήταν πολύ σαφή τα σχόλια και ευχαριστώ για τη συμφωνία που έδειξε ότι αφορά την μετανομασία των αποστολών σε επισκέψεις διαλόγου. Σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα, εύστοχο είναι το σχόλιο σας σε ό,τι αφορά την προσδιορισμό του προστήμου καταρχήν σε ένα αποθεματικό και μετά σε πραγματική επιβολή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μία τέτοια πρόταση θα μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε εφόσον συγκεκριμενοποιηθεί σε μια τροπολογία ή συμβαστική τροπολογία. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και το πού θα αποδίδονται, η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών προβλέπει ότι τα πρόστιμα περιέρχονται στο μηχανισμό σταθερότητας. Αντιλαμβάνομαι ε, τη μάχη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιέρχονται τα πρόστιμα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εγώ πάντως ε, προσπαθώ να εφαρμόσω αυτή την καρτισιανή προσέγγιση, όπως σας είπα στην αρχή. Δηλαδή, ο κανονισμός αυτός να είναι όσο πιο παράλληλος γίνεται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως είχαμε συμφωνήσει άλλωστε. Σας ευχαριστώ. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση ΕΠΕΝΚ λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου. Θα τη συζητήσουμε στις 23 Ιανουαρίου, προκειμένου να ψηφίσουμε στις 12 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Αυτό είναι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Τις αφήνω για αργότερα όταν έρθουν οι συνάδελφοι για την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 9.40 ε, και 50. Ε, Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα λοιπόν μέχρι ότου έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Could you, could you take your seat? Παρακαλώ συνάδελφε καθίστε. Thank, thank you very much. Um, I'll proceed now as usual with the... Θα περάσουμε πρώτα στις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Δύο ανακοινώσεις έχω. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα δεν θα ψηφίσουμε ε, μία από τις εκθέσεις που προβλέπονται. Επίσης, έχει ε, συμφωνηθεί υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου και υποβολής εκθέσεων. Για την περίοδο 2014-2020 ήταν ο τρίτος τριμερής διάλογος και στις 3 Δεκεμβρίου καταλήξαμε σε συμφωνία για το μελλοντικό χρηματοδοτικό σύστημα υποστήριξη τρεις ε, οργανώσεις ε, στον τομέα Τη υποβολή εκθέσεων και δημοσιονομικού ελέγχου ΕΦΡΑΚ, ISP και PIOB. Θα γίνει νέα διαβούλευση με την Επιτροπή μας ε, στις 9 Δεκεμβρίου. Χθες είχαμε και τον 10ο ε, πολιτικό τριμέρι διάλογο για τη ΜΥΦΙΤ. 7 ώρη διάρκεια. Σε αυτό το παγωμένη, σε την παγωμένη αίθουσα δεν αισθανόμουν τα πόδια μου στο τέλος. Είχα μου διάσει, αλλά ευτυχώς είδα ότι σήμερα ε, το έχουν φροντίσει. Έχουμε συμφωνήσει για τη διάρθρωση της αγοράς, προχωρούμε στο θέμα των τρίτων χωρών, τώρα για τα, για, τα εμπορεύματα και την πρόσβαση στις αγορές έχουμε ακόμη δρόμο. Έχουμε πάντως ε, πρόγραμμα και, την, και για την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτο θα ψηφίσουμε τον ορισμό στη θέση του Πρόεδρου του Εποπτικού Συμβούλου της κυρίας Δανιέλ Νούι. Ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο πρώτα αν έχετε, λάβει, αν έχετε μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας. Γίνεται δοκιμαστική ψηφοφορία για να ελέγξουμε πρώτα τις συσκευές. Anybody 31 members είναι παρόντες, 24 ψήφισαν υπέρ. Ωραία, λειτουργούν τα μηχανήματα. Ψηφίζουμε την έκθεση της Προέδρου, παράγραφος 1, αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τη λογική σκέψη 1 προς 5 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α προς ε, τη λογική σκέψη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 29 ψήφισαν υπέρ, κανείς κατά και μία αποχή. Οπότε εγκρίνεται ο ορισμός, θα παραπευθεί το θέμα στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας. Τα κέρματα δεν θα τα ψηφίσουμε. Και προχωρούμε, το 5 επαναλαμβάνω αναβάλλεται, τα κέρματα αναβάλλονται. 6. Ενιαίοι κανόνες και ενιαία διαδικασία. Ε, και αυτό αναβάλλεται ε, για τις 17 Δεκεμβρίου. Α, και έληξε η ψηφοφορία.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 Um, Θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 7, έκθεση της Προέδρου για τους ε, δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις. Ήδη είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Θα θυμάστε ότι σας είχα μοιράσει εγκαίρως ε, ένα σχέδιο έκθεσης Έγινε μια επικαιροποίηση στο μεταξύ. Διευκρινίστηκαν κάποιες λεπτομέρειες. Θα περιμένω να αποκατασταθεί η ησυχία στην αίθουσα και μετά θα συνεχίσω. So those, those leaving can do so quietly, please. Παρακαλώ όσοι φεύγουν να, το κάνουν χωρίς φασαρία είπα λοιπόν, έγινε μια ενημέρωση της, του πρώτου σχέδιου που σας είχα μοιράσει. Διευκρινίστηκαν κάποιες λεπτομέρειες και έκτοτε είχα συζητήσεις με πολλούς συναδέλφους και άκουσα πολλά σχόλια για ειδικά είδη δικτών αναφοράς. Και φρόντισε αρκετά το κείμενο. Το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά ήταν ευρύ, κάλυπτε όλους τους δείκτες ε, ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς για την ε, απόδοση μιας, ε, ενός ταμείου επενδυτικού ή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή Εγώ καθο... περιόρισα περισσότερο στους διαχειριστές ε, των δικτών ε, το κείμενό μου. Και μάλιστα όταν ένα δείκτη αναφοράς εμπίπτει σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε θεωρώ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Με αυτή τη βάση έκρινα ότι αν δίνουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να είναι αυτοί αξιόπιστοι. Δεν περιορίζεται σε κρίσιμους δείκτες αναφοράς όπως το LIBOR και το EURIBOR. Είναι κάπως πιο ευρύ το πεδίο εφαρμογής. Επίσης ε, ρυθμίζουμε και τους οίκους αξιολόγησης, τη μεθοδολογία και τις αρχές και όχι τις αξιολογήσεις καθ' αυτές. Έχω καταθέσει και αρκετές τροπολογίες για να λάβω υπόψη το θέμα της αναλογικότητας. Αυτό γίνεται σε διάφορες φάσεις και στους κανόνες της ε, ΕΣΜΑ, της ΕΑΚΑ και σε τη φορά την αίτηση αδειοδότησης. Οι αρμόδιες αρχές ε, μπορούν στη φάση αυτή να αποδείξουν αν ένας διαχειριστής ευθύνεται για περισσότερους δείκτες αναφοράς και αν ε, χρειάζεται αναλογική μεταχείριση. Σε μεταγενέστερο στάδιο αυτό αποφασίζεται. Επίσης προβλέπω ότι ουσιαστικά κάθε δείκτης αναφοράς ε, ε, που μπορεί να δημιουργεί ανησυχία μπορεί να περιληφθεί στον κανονισμό. Επίσης, όταν μια οργάνωση διαχειριστής αποφασίζει ότι ένας δείκτης αναφοράς δεν αξίζει να εμπίπτει στον κανονισμό, μπορεί να αφαιρεθεί. Αυτό όμως γίνεται από υποβολή αίτηση στις αρμόδιες αρχές, γιατί αυτές ε, το κρίνουν. Και σε ό,τι αφορά την αφαίρεση του δικτύου αναφοράς υπάρχουν ε, τεχνικές προδιαγραφές ε, και νομοθετικές που θα πρέπει να τηρηθούν. Άρθρο 5 που μιλάει για τον ρόλο της ΕΚΑ, της ΕΣΜΑ. Είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος και δείχνει πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία με τις κατευθυντήρες γραμμές και τις ε, τεχνικές και ρυθμιστικές προδιαγραφές. Στο πρώτο επίπεδο δεν ε, ε, ξέρεις αυτόματα τις κεντρικές τράπεζες, αλλά ανέφερα παρακάτω τους αξιωματούχους για στατιστικά θέματα που μιλούν που σχολιάζουν τις οργανώσεις που υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο και για το κατά πόσο εμπίπτουν στις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΑΚΑ. Μπορεί η ΕΑΚΑ, αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ε, να, να αφαιρέσει κάποιες συναλλαγές από τις διατάξεις. Ίσως ε, αυτή η προϋπόθεση τροποποιηθεί ανοίγοντάς την περισσότερο στην αναλογικότητα. Να μην έχουμε μόνο απλώς εισαγωγή αφαίρεση, αλλά λήψη υπόψη της αναλογικότητας. Γιατί ίσως κάποια στοιχεία του κανονισμού δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν αν κάποιες ε, πληροφορίες είναι δημοσίως προσιτές. Πιστεύω πάντως ότι οι αρμόδιες αρχές και η ΑΚΑ θα κατακλειστούν από τον τεράστιο όγκο των δικτών αναφοράς και των διαχειριστών και ίσως θα απελαγώσουν στην αρχή. Γι' αυτό καλό θα ήταν να προτείνουμε μια σταδιακή εισαγωγή. Όπως, όπως έγινε και με τα παράγωγα και θεωρήσαμε ότι είναι αδύνατον από την αρχή αμέσως να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού. Υπήρχε λοιπόν μια σταδιακή, σταδιακή εισαγωγή με τα πιο σημαντικά πρώτα και μια ιεράρχηση. Μια τέτοιου είδου ιεράρχηση θα πρέπει ίσως να γίνει και τώρα για να μην πελαγώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών οι αρμόδιε αρχές. Και αυτή την αρχή πρότεινα στο, στο τέλος του άρθρου 5 και τη θεωρώ πολύ σημαντική. Επίσης την ΕΑΚΑ την έβαλα και σε άλλα σημεία. Ίσως θα πρέπει να εκχωρηθούν και, άλλες, και άλλα καθήκοντα και περιμένω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Άλλο μείζον θέμα είναι οι διατάξεις για τις τρίτες χώρες. Της τροποποίησα ώστε να αντανακλούν η ρύθμιση διαχειριστών χρηματοπιστωτικών δικτών αναφοράς είναι σε μεγάλο βαθμό μια εξελισσόμενη διαδικασία. Πολλές τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να ρυθμίσουν τους δείκτες αναφοράς ή άλλους δείκτες με βάση τα πρότυπα της ε, ΙΟΣΚΟ, όπως είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ίσως δημιουργηθεί και πρόβλημα για τις ισοδυναμίες των τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δούμε αν είναι ισοδύναμη η νομοθεσία ή αν θα καθυστερήσει μια τέτοια ισοδύναμη νομοθεσία. Οπότε προβλέπονται και εδώ δύο στάδια σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ΑΙΟΣΚΟ. Πρότεινα μια μεταβατική περίοδο που είναι ε, 13 μήνες, 30 μήνες συγγνώμη, είναι κάπως ε, πιο μακρά. Η ε, διαδικασία διαδικασίες της πρώτης φάσης, δηλαδή πριν την αναθεώρηση, δύο έτη πιστεύω πριν ε, υποβληθεί το αίτημα αδειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ήταν σκόπιμο λοιπόν να δώσουμε αυτούς τους 30 μήνες στις τρίτες χώρες. Επίσης, ε, ό,τι οι διαδικασίες σταδιακής αγωγής ε, προτείνουμε θα ισχύσουν και για τις τρίτες χώρες. Ίσως ε, δεν λειτουργεί στο σύστημα πλήρως και ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε πιο ευρηματικές λύσεις σαν αυτή που αναφέρουμε στο Omnibus 2 για τις Ηνωμένε Πολιτείες όταν δεν υπήρχαν ισοδυναμίες. Γιατί δεν υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ασφαλίσεις, οπότε προβλέψαμε κάποιες ε, προσωρινές ισοδυναμίες. Κάτι τέτοιο ίσως προτείνω και εδώ για τις τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση για τις τρίτες χώρες, θεωρώ ότι η εποπτική αρχή που θα χρησιμοποιήσει τους δείκτες αναφοράς να προτείνει κάποια τα τεκμήρια, κάποιες αποδείξεις που να τεκμηριώνουν συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ΙΟΣΚΟ. Έτσι θα στοιχειοθετείται ισοδυναμία. Αυτές οι πληροφορίες θα μεταβιβάζονται στην αρμόδια αρχή και στην ΕΑΚΑ. Έτσι θα μπορέσει η ΕΑΚΑ να καταρτήσει τον ασφαλή κατάλογο, όπως λέμε, safe list. Οπότε αυτός ο κατάλογος θα λαμβάνεται υπόψη και από για να βλέπουν ότι κάποιος διαχειριστής δίκτυα αναφοράς ή ένας συγκεκριμένος δίκτυας αναφοράς έχει ήδη εγκριθεί. Και θα μπορεί ο κλάδος να συμβουλεύεται αυτό τον κατάλογο και να βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές. Ε, περιμένω τις ιδέες σας και τις συστάσεις σας για τα σημεία αυτά, αλλά πραγματικά εγώ δεν βρήκα άλλο τρόπο ισοδυναμίας γιατί δεν ήταν επίσημο αυτό το θέμα της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της ΙΟΣΚΟ. Τώρα, διαφάνεια. Η διαφάνεια των δεδομένων και των μεθοδολογιών που εφαρμόζεται για την παραγωγή δίκτυα αναφορά είναι χρήσιμο εργαλείο για του επενδυτέ και τι εποπτικέ αρχέ. Άλλοι ε, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και τις μεθοδολογίες. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μία νέα λύση για όλους και για τους δείκτες αναφοράς. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή για σημαντικές επενδύσεις, αυτοί θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μετά από συγκεκριμένη περίοδο. Και υιοθέτησα αυτή τη διατύπωση, γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με τέτοιου είδους δεδομένα αν ε, υπάρχει μια άδεια για την οποία έχει καταβληθεί τίμημα και θέλουμε ε, άμεσα από τις ε, συναλλαγές να καταλαμβάνετε και ένα τίμημα, να καταβάλλετε και ένα τίμημα. Μετά από λίγο καιρό όμως ούτως ή άλλως δημοσιοποιείται. Οπότε αναγνωρίζουμε τα εμπορικά συμφέροντα που υπάρχουν και προβλέπουμε την απαραίτητη διαφάνεια περιμένοντας να την περίοδο ώστε να δημοσιευθούν, να δημοσιοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Γιατί είναι σημαντικό να ελέγχονται, να ελέγχεται η παραγωγή των δικτών αναφοράς και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν. Σε ό,τι αφορά τα εισερχόμενα δεδομένα και τη μεθοδολογία, άλλαξε κάπως ε, το κριτήριο της διαφάνειας και είπε ότι σε κάποιο στάδιο μιλούμε για δημοσίευση του, είτε του δεδομένου είτε της μεθοδολογίας όταν μιλάμε για διαφορετικά μοντέλα. I think point talk about... Το τελευταίο σημείο θα το διαβάσετε και στην έκθεση, αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πάυση παροχής δίκτυα αναφοράς εφόσον ε, θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό ανέφερα και τη διάταξη για τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς. Αν ε, δεν είναι αρκετοί αυτοί που συμβάλλουν, ίσως ε, θα μπορούσαν υποχρεωτικά να θεσπίσουμε τη συμβολή. Η, ΕΣΚΑ, η ΕΑΚΑ συγγνώμη, πρέπει να ενημερώνει τους, δια, διαχειριστές, να διαβουλεύεται μαζί τους και να καταβάλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να ακολουθεί τις αρχές της ΙΟΣΚΟ. Κατά του τελευταίου μήνε έχει επίση παρατηρηθεί σταθερή μείωση τη υποβολή ερχόμενων δεδομένων για το Libor και, το Euribor και το 20% κατόφλι από την Επιτροπή για την ενεργοποίηση αυτής της απέτηση για την υποχρέωση δηλαδή συμβολής δεν είναι αρκετά ελαστική. Για το Euribor για παράδειγμα, αν δεν έχουμε καμία συμβολή από ένα κρατος μέλος ή από μια ομάδα κρατών μελών, αυτό δεν θα πρέπει κατά ανάγκη να ενεργοποιεί το, το όριο του 20%. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στην πρόταση της Επιτροπής. Γιατί μερικές φορές δεν υπάρχουν ε, αρκετές πληροφορίες. Ίσως θα πρέπει και εδώ να ενισχύσουμε το ρόλο της ΕΑΚΑ. ώστε όταν απαιτείται μία πληροφορία να εξασφαλιστεί η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το για, τα τέλη και την αδειοδότηση και εδώ με ενδιαφέρει η διαφάνεια στην, στον υπολογισμό και στη διάρθρωση των τελών, ώστε να μην ε, γίνεται αθέμητη επιδότηση ουσιαστικά και να μην να γνωρίζουν οι, οι ενδιαφερόμενοι αν υπάρχουν τέλη ε, ενσωματωμένα στους δείκτες αναφοράς. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια της μεθοδολογίας και των εισερχόμενων δεδομένων, η ΑΚΑ θα πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα διαλύματα ε, για και το χρόνο στον οποίο θα δημοσιοποιούνται αυτά. Θα δούμε τι διατύπωση θα βρούμε για το σημείο αυτό. Αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη επισκόπηση της έκθεσής μου. Θα ακούσουμε τώρα τους και ηγητές. Ο Γκέι Μίτσελ πρώτος από το ΕΛΚ. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την λεπτομερή εισήγηση που την οποία συμμερίζομαι, συμμερίζομαι και τις ανησυχίες σας. Ε, κινούμεθα με ταχύτητα φωτός, μας ε, προλάβατε λίγο ε, εσύ και σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω πως εν γέννη μπορούμε να βρούμε μια γενική συμφωνία για πολλά από τα σημεία που αναφέρατε. Δεν είχα την ευκαιρία ωστόσο να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου του ΕΛΚΑ αλλά θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμή. Για το θέμα του πεδίου εφαρμογή, σα ευχαριστώ για τι προτάσει περί επέκταση του πεδίου. Εγώ καλωσορίζω τις προσπάθειές σας για κατηγοριοποίηση των διαφόρων ε, οροσίμων. Ε, περιμένω να με πείσετε, αλλά φοβούμαι πως η χρήση ε, οροσίμων που μπορεί να αλλάζουν διαχρονικά μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Αλλά, με περιπτώσει, πρόκειται για μια ευκαιρία για να συζητήσουμε για τους δείκτες αυτούς αναφοράς. Εγώ θα πρότεινα να αφαιρέσουμε το κατόφλι των 100 δις και να το τοποθετήσουμε με διαφορετική διατύπωση επί τη βάση του αντικτύπου στους καταναλωτές και της δυνατότητας να απειλήσουν την ακυρεότητα της αγοράς και όχι με βάση τον ίδιο τον όγκο. Και αυτό θα μπορούσε να υπόκειται στα αριθμιστικά πρότυπα, ε, όπως ε, λέει και η τροπολογία 37 της εισηγητρίας και ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και μια διάταξη ώστε η Κομισιόν να μπορεί να υιοθετεί εφαρμοστικές πράξεις για την εφαρμογή δικτών αναφοράς καθώς και κρίσιμων δικτών αναφοράς και να δίνεται έτσι περισσότερο ε, περιθώριο στους ε, ρυθμιστές ανάλογα με το αν οι δείκτες αναφοράς είναι πιο προβληματική ή όχι. Αυτό ήθελα να το τονίσω και όπως είπα και στην αρχική μας συνεδρίαση νομίζω πως αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις κεντρικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και ελπίζω να βρούμε συμφωνία γιατί αυτοί, ε, αυτές ε, είναι αντικείμενο εποπτείας από πλευρά της Eurostat και ήδη υπόκειται σε αυτή ε, πρότυπα και προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια ε, και δεν θεωρώ πως είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν λοιπόν στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Όσον αφορά το κώδικα διοντολογίας ε, των ε, συμβαλλόντων και ιδιαίτερα σε σχέση με το άρθρο 9, εδώ υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται για τον κώδικα διοντολογίας θα πρέπει να σκεφτούμε την εξή διατύπωση για το άρθρο 9.2. Για το κώδικα ζητολογίας θα πρέπει να υπογράφεται από το διαχειριστή και από του ε, ε, συνεισφέροντε και θα είναι δεσμευτικά, νομικά, νομικά δεσμευτικό από τη στιγμή που αυτό είναι πρακτικό και ο διαχειριστή θα πρέπει να αποδείξει πω ε, αυτό ο κώδικα ζητολογίας ισχύει, αλλά ότι έχουν γίνει αποκλήσει από τη στιγμή που δεν γινόταν να εφαρμοστεί. Αυτή είναι μια πρώτη απόπειρα για νέα διατύπωση. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε κάποια ε, συμφωνία για τη διατύπωση. Όσον αφορά τώρα τους διαχειριστές ε, περιουσιακών στοιχείων, ε, ο στόχος είναι να μην είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές ε, των στατιστικών στοιχείων και η τροπολογία 55 της συγκεκριτηρίας μπορεί να είναι βελτίωση, φαίνεται να είναι βελτίωση και η διαγραφή της λέξης εμπορεύσιμο στην, στην ε, τροπολογία της εισηγήτριας νομίζω πως θα ε, ακόμη περισσότερο την ε, συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφερθήκατε επίσης ε, στα καθεστώτα τρίτων χωρών ε, και είμαι γενικά υπέρ, αλλά γνωρίζω πως υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες που δεν φανίζονται αυτή τη στιγμή, ώστε να, να, κάνουμε βήματα για να εφαρμοστούν οι αρχές της ΕΚΑ τη ΣΥΟΣΚΟ. Ε, νομίζω πως θα, καλό θα ήταν να ενισχυθούν οι προτάσεις σας μέσω ε, να ενισχυθούν οι προτάσεις μάλλον για τους διαχειριστές τρίτων χωρών που θέλουν να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες αναφοράς τους στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προβαίνουν σε δήλωση ε, που θα υποβάλλεται στην ΙΟΣΚΟ. και θα προβλέψουμε και κυρώσεις αν αυτές οι δηλώσεις είναι ψευδείς, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των διαχειριστών τρίτων χωρών στις, στην αγορά μας. Για, το θέμα των σχετικών στοιχείων δεν έχω πρόβλημα. Ε, μάλλον μου έχουν γνωστοποιήσει τα χρηματιστήρια ότι το θέμα έτσι όπως έχει ε, συμπεριλαμβάνει στοιχεία και από αριθμιστικά σώματα Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αριθμιστικά στοιχεία και τα στοιχεία OTC, over the counter. Ε, Υπάρχει και το θέμα των πληροφοριοδοτών και ως προς αυτό άκουσα διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και κανείς δεν είχε αντίρρηση για την ενίσχυση των διατάξεων περί ε, πληροφοριοδοτών και μάλιστα τις διατάξεις ε, του, του ΜΑΡ που ζητούν ίσως και χωριστές ε, σχετικές διατάξεις. Δεν είμαι βέβαιος ακόμα, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να εισάγουμε μια χωριστή διάταξη. Τώρα για το άρθρο 24, δηλαδή τα σύνολα αρμόδιων αρχών. Εδώ ακόμα δεν είμαι βέβαιος, ε, νομίζω πως θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Εγώ πιστεύω πως κάνατε εξαιρετική δουλειά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ελπίζω πως θα ανταποκριθούμε στο χρονικό πλαίσιο για το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό αυτό ώστε να έχουμε τελικά έναν καλό κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Γκέιν. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Έμιλη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ Πρόεδρε και για τη δουλειά σας, για την ε, έκθεση την οποία καλωσορίζουμε. Μας άρεσε βέβαια και η έκθεση τη Επιτροπής, αλλά βλέπουμε ότι βελτιώνεται σε το κείμενο αναζητώντας κάποιες λύσεις. Ε, νομίζω βέβαια ότι χρειάζεται να συστήσουμε ακόμη περισσότερο κάποια πράγματα. Πάντως, εν γέννη, μας ενδιαφέρει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτό το ζήτημα της αυτορύθμισης για τους δείκτες αναφοράς. Αυτά που είδαμε από τις υποθέσεις ε, τις περσινές αλλά και στην, ε, στις ανταλλαγές, ε, στις συναλλαγές σε βασικά αγαθά ή στις προδιαγραφές για τον χρυσό, αντίστοιχε δηλαδή περιπτώσεις, ε, είναι ότι χρειάζεται ρύθμιση. Και φαντάζομαι ότι και εσείς τα ίδια μελήματα, και εσάς τα ίδια μελήματα σας κινούν. Ε, γι' αυτό μιλάμε για ένα πεδίο αναφορά στο δυνατόν πιο ευρύ. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα αποκλειστεί από το πεδίο ή τι δεν θα περιλάβουμε στο πεδίο αναφοράς γιατί εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα, ε, αυτές οι αγορές και πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο προσεκτικοί. Στο τι θα ρυθμίσουμε βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε όπως προτείνετε και εσείς να υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή. Στην υποχρεωτική συνεισφορά για τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς, στο άρθρο 14 δηλαδή, συμφορούμε με την τροπολογία σας, την 63, ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και από τις, ε, από τις ε, αρχές διαχείρισης να δημοσιεύουν τα στοιχεία για την εταιρεία και τους δείκτες και επίσης περισσότερη ευελιξία που ζητάτε για την υποχρεωτική συνεισφορά το 23 δηλαδή που αναφέρεται και εμείς θα συμφωνήσουμε και Το όριο 20%. Επίσης, στην 101 τροπολογία συμφωνούμε, συμφωνούμε με τις ανησυχίες σας ότι μπορεί να είναι κάπως ε, περίπλοκο το ζήτημα και ότι χρειάζεται μια κάποια διευκρίνηση διατύπωση. Θα συμφωνήσουμε με εσάς. Για τους πληροφοριοδότες whistleblowers έχετε δεχθεί τις προτάσεις. Βλέπουμε στην ε, τροπολογία 59 και το άρθρο 11, συμφωνούμε. ευθύνες αρχών διαχείρισης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των διαχειριστών. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωστόσο θα πρέπει πιστεύω ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση και να πιέσουμε και τους συνεισφέροντες περισσότερο από ό,τι τώρα. Ένα παράδειγμα. Όταν συζητήσαμε το Τάιμπερ στην ε, Δανία, την, το διατραπεζικό επιτόκιο, το διαχειριζόταν η Κεντρική Τράπεζα, η οποία παρετήθηκε όμως το 2007, μας λέει δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τι συμβαίνει, να διαφανίσει η διαδικασία, δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητα των συνεισφορών. Και ως εκ του ε, απεκδίωμαστε τις ευθύνες. Βεβαίως μπορούν να έχουν την απέτηση να απαιτήσουν δηλαδή πληροφορίες από το συνεισφέροντα και ως ε, διαχειριστές μπορούν να διατυπώσουν απαιτήσει προς τους ε, συνεισφέροντες, αλλά η, το παράδειγμα σας το, δείχνω, σας το δίνω για να δείξω πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η δουλειά των ε, διαχειριστών και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ε, δουν ξεκάθαρα την εικόνα του τι συμβαίνει. Αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τροπολογία εκεί. Ένα προβληματισμό ήθελα πως τώρα να εκφράσω και την ανάγκη να το σκεφτούμε καλύτερα. Το συλλογικό όργανο της αρμόδιας αρχής στην τροπολογία, στις τροπολογίες 104-108 έχουμε κάποιες επιφυλάξεις γιατί βλέπω ότι το συλλογικό αυτό όργανο το μετατρέπει σε ένα όργανο συλλογή πληροφοριών, άρα αποδυναμώνεται ο ρόλο του σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή, όπου έχει αποφασιστικό ρόλο και σίγουρα ε, σε σχέση με την πρώτη, απόφαση, με την πρώτη πρόταση της Επιτροπής που τιμούμε εμείς. Γι' αυτό θέλουμε πιο ισχυρό ρόλο του συλλογικού ε, οργάνου εάν μιλούμε για δείκτες αναφορά, της, αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον είναι κάτι το τόσο σημαντικό πρέπει να έχει και η ΕΣΜΑ τους ε, ε, τον καθοριστικό ρόλο. Για τις κυρώσεις πρέπει να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο σχέση με τη Market CRD4. Θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα ποιο είναι το, το κρινόμενο ζήτημα, διακυβέρνηση ασφαλώς και η απευθείας επέμβαση, κατάχρηση δηλαδή στην αγορά, το οποίο είναι ένα ζήτημα, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το επίπεδο παρέμβαση το οποίο σκοπεύει να προτείνει, που, είναι, που έχει προτείνει μάλλον γιατί είναι χαμηλότερο από αυτό της κατάχρηση τη αγορά. το οποίο των κυρώσεων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να μα εξηγήσουν γιατί. Για εδώ τον κώδικα συμπεριφορά που σχετίζεται βέβαια και με τι τρίτε χώρε, και το όλο αυτό ζήτημα, το οποίο κρίνω πιο δύσκολο ασφαλώς. Γιατί θέλουμε βέβαια να θέσουμε ε, προδιαγραφές ποιότητας εμείς, αλλά πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και το σύστημα. Και ένα άλλο ζήτημα. Θα πρέπει ε, ο κώδικας συμπεριφοράς να είναι δεσμευτικός νομικά. Σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα και γι' αυτό θα ήθελα να το κοιτάξω λίγο πιο προσεκτικά για να διατυπώσουμε μια πιο συγκεκριμένη θέση. Γιατί βλέπω κάποια ζητήματα που με προβληματίζουν. Εν όλο, καλή δουλειά σας, σας ευχαριστούμε πολύ και με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ, Έμιλι. Ο Φιλίπ Λάμπερτ, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Και εγώ μπορώ να συμμεριστώ πολλά από αυτά τα οποία είπαν και οι τρει προλαλήσαντε. Άρα βλέπω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Σε κάποια θέματα μόνο θα επικεντρωθώ. Οι δύο οι στους οποίους δεν είμαστε 100% βέβαιοι για τις επιλογές, για τις προτιμήσεις μας, είναι το καθεστώς ή διατάξεις ειδικές με τις χώρες, τρίτες χώρες και το ζήτημα του περιορισμού του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού να απευθύνεται δηλαδή στους διαχειριστές ε, δίκτωρων αναφοράς. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι... Βεβαίως είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι είναι και ο πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό που έχει επιλεγεί. Είμαστε ακόμα αναποφάσιστοι. Για τους ορισμούς και το πεδίο αναφοράς. Θα περιλαμβάναμε και τα χρηματοπιστωτικά μέσα OTC of the country, με διαγραφή δηλαδή του άρθρου 3 παράγραφος 15. Θα έσαγαγαμε έναν ε, ορισμό των ε, δικτών αναφορά ξέρου συναλλάγματο και θα μειώναμε το όριο για τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς. Θα ε, ήθελα δεν να επιμείνω και σε αυτό ίσως να έχουμε αποκλίνουσα θέση, με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες ομάδες και με την Επιτροπή και την πρότασή της. Πιστεύουμε ότι τα επιτόκια και οι δείκτες αναφοράς ξένου συναλλάγματος θα πρέπει να βρίσκονται στην άμεση εποπτεία της ΕΣΜΑ. Αυτό άλλωστε δείχνει και ο ρόλος της στον έλεγχο της ιστορικής αγοράς. Δεν βλέπω γιατί δεν θα πρέπει να έχει αυτή την ευθύνη η ΕΣΜΑ. Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΣΜΑ στα συλλογικά όργανα για τον προσδιορισμό των δικτύων αναφοράς. Όπως υπόθηκε και νωρίτερα, εάν θέλουμε με σοβαρότητα να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να τον αλάβει η ΕΣΜΑ, ε, γιατί έχουμε να κάνουμε με, ένα πανευρωπαϊ... με πανευρωπαϊκές αγορές και ίσως και παγκόσμιες και γι' αυτό ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η ΕΣΜΑ. Οτιδήποτε λοιπόν αποκλίνει ή ξεφεύγει από τον έλεγχο της ΕΣΜΑ θα πρέπει να καλυφθεί από μια ρήτρα αναθεώρησης που θα λέει ότι τίνουμε προς, το, προς την τροποποίηση στο σκοπό αυτό, στο μέλλον. για το ρόλο της. Δεν ξέρω γιατί η Επιτροπή έχει κάνει τις επιλογές αυτές, αλλά πάντως ε, έχουμε μια εσωτερική αγορά η οποία βλέπουμε να μην λειτουργεί ικανοποιητικά ε, και σε αυτό θα πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα. οι διεθνείς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να ρυθμίζονται σε διεθνές επίπεδο εν τέλει. Ευχαριστώ. Κύριε Σέπιν, εκ μέρου της CCR. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Σαΐτ Καμέλ. Ε, είναι πρόσδεκτη η έκθεσή σα. Αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με αυτά που αρχικά είχε προτείνει η Επιτροπή. Όσον αφορά το πεδίο αναφορά, με χαρά διαπιστώνω ότι η να περιορίσει το αποφάσισε να περιορίσει το πεδίο αναφορά προ τη συστημική χρήσιμα στοιχεία του. Ε, δεν συμφωνώ 100% με τα όσα έχετε συμπεριλάβει ωστόσο, ιδιαίτερα το αυθαίρετο ποσό των 100 ευρώ. Νομίζω ότι όμως συμφωνούμε επί της αρχής. Δεν πρέπει να λησμονούμε γιατί υιοθετήθηκε αυτός, αυτή η πρόταση. Δηλαδή ότι σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει διαπιστώθηκαν αδυναμίε και πρέπει να εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωση του κανονισμού το χειτερό δυνατό. Πράγμα το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε εάν. Ε, τακτοποιήσουμε τα τον Άιμπορ και αφήσουμε τους τίτες αναφοράς να, τεθούν σε, να ενταχθούν στο σύστημα αργότερα. Πρέπει να προσέξουμε να μην βρεθούν σε σύγκρουση κίνδυνοι για τον καταναλωτή και με τους συστημικούς ε, κινδύνους. Θα ήταν εσφαλμένο να παραγνωρίσουμε αυτό το κίνδυνο και πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο ευέλικτο καθεστώς. Κάθε κράτος, κάθε μεγάλη οικονομία θα πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην υιοθέτηση των αρχών ΙΟΣΚΟ, γι' αυτό δεν θα πρέπει εμείς να αυτοαπομονωθούμε. Τα πράγματα βαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση, κυρία Πρόεδρε, και αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την στέοχευση του, του κανονισμού στα, στους δείκτες αναφοράς, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να κλείσουμε το θέμα αυτό. Κυρία Μπόλς, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση. Μια στιγμή, γιατί έχω κατάλογα. Ο Βέρνερ και μετά ο Όλαφ. Βέρνερ. Συγγνώμη, ε, λησμόνησε έναν σκιώδη γιατί δεν τον είχα στον κατάλογο. Μίαν σκιώδη. Δεν ενημερώθηκα. Επιστρέφω λοιπόν. Γκούε. Σα ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ε, ε. Για την πρόταση ακούσαμε πάρα πολλά σχόλια. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο από τη δική μου πλευρά, αλλά όπως και ο Φιλίπ και όπως, ε, όπως και οι άλλοι προελίσσαντες, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα, μεγάλη δυνατότητα και πολλές ελπίδες να καταλήξουμε στη συμφωνία. Γιατί επί της ουσίας δεν έχουμε προβλήματα με την πρόταση της συγκήτριας. Υπάρχει ευρία βάση για τη συνένεση μεταξύ μας λοιπόν και ιδιαίτερα σε, σε κάποια σημεία έχουμε απόλυτη σύμπνοια. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ε, ε, αλλαγές στους δείκτες αναφοράς και τις εξουσίες των εποπτικών αρχών. Επίσης, ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής ε, και τον περιορισμό του και εμείς ε, στενιζόμαστε τις ανησυχίες κάποιων συναδέλφων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να δούμε τι εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογή. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται ένα κατάλογο ε, με του δείκτε αναφορά ε, που εμπίπτουν στον κανονισμό, θα πρέπει να προσέξουμε τι αφήνουμε απ' έξω. Συμφωνούμε με την αναλογικότητα και συμφωνούμε με την πρόταση για την ΕΣΜΑ, την ΕΑΚΑ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Θα πρέπει όμως να δούμε τι είναι εφικτό. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας και Έρευνας, έχω κάποια προβλήματα. Μερικά αφορούν τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και άλλα αφορούν την έκθεση την ίδια. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, τα commodities, έχουμε πρόβλημα γιατί έχω την αίσθηση ότι εμείς ε, προσπαθούμε να μην ε, δημιουργήσουμε ένα, ε, ένα χάος που δεν θα μπορούμε να το ρυθμίσουμε γιατί υπάρχουν διεθνείς κανόνες και διεθνείς προδιαγραφές από την ΙΟΣΚΟ που αφορούν τα προϊόντα και έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες τη διαδικασία αξιολόγησης, για παράδειγμα, αυτών των ε, κανόνων. Και μάλιστα η αξιολόγηση αναμένεται για τον Απρίλιο του 2014. Συμπίπτει δηλαδή με τη δική μας ε, εξέταση της πρότασης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, αυτά τα συστήματα θα συστηθούν εκ παραλίλου. Δηλαδή, αφενός η δική μας πρόταση, αφετέρου η αξιολόγηση που θα ολοκληρωθεί από την ΙΟΣΚΟ. Και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις ως προς τη γενική πρόταση, συμφωνώ με τη Σάρων Μπόλς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τριαντάμινη μεταβατική περίοδο. Συμφωνώ με τη μεταβατική περίοδο και με τη διεύρυνσή της στους 30 ε, μήνες. Τώρα για τα προϊόντα, ίσως η συζήτηση θα πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος και ίσως παρουσία και των σχεδόν εισηγητών της Επιτροπής Ήτρε. Υπάρχουν τρία προβλήματα που δεν έτυχαν της δέουσες ε, εμβάθυσης και ανάλυσης. Και παρόλα αυτά είναι σημαντικά και δεν μπορούν να γνωριθούν. Φοβάμαι ότι ίσως με τις νέες απαιτήσει μειωθούν οι συνεισφορές ε, και υποβαθμιστεί η ποιότητα των δικτών αναφοράς. Ένα τέτοιο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, θα επιληθεί μόνο με την αύξηση των ε, εξουσιών των διαχειριστών. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αφορά το γεγονός ότι οι δείκτες αναφοράς ε, επιδέχονται και εξέλιξης και αντικατάστασης, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση ε, των δικτών αναφοράς που περιλαμβάνονται σε μακροχρόνιες συμβάσεις για να μην χαθεί αυτή η έννοια της, του σημείου αναφοράς που εξασφαλίζουν αυτοί οι δείκτες. Τρίτο σημαντικό πρόβλημα της γενικής πρότασης αφορά τις αλλαγές στη μεθοδολογία. Πιστεύω θα πρέπει να ελέγχονται αυτές οι αλλαγές ε, στις μεθοδολογίες και θα πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε μια αλλαγή της μεθοδολογίας να χρησιμοποιηθεί ως ε, εργαλείο παραποίησης ή χειραγώγησης ή κατάχρησης. Αυτά είναι τα τρία γενικά προβλήματα, γιατί οι συνάδελφοι κάλυψαν περισσότερα τα ειδικά προβλήματα. Επίσης, ε, το θέμα των διοικητικών ε, κυρώσεων. Γιατί στην παράγραφο 31, στο άρθρο 31, στη δεύτερη παράγραφο, εκεί που μιλούμε για τις προσωρινές απαγορεύσεις κατά ιδιωτών που έχουν κατηγορηθεί για, για παραβιάσεις, γιατί στις εξαιρέσεις περιλαμβάνουμε μόνο κάποιες διοικητικές λειτουργίες. Δεν θα πρέπει να περιορίζομαστε μόνο στις διοικητικές λειτουργίες, θα πρέπει να μιλούμε γενικότερα για λειτουργίες στην περίπτωση των προσωρινών εξαιρέσεων. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο γενικό κατάλογο των ομιλητών. Ο Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τόσο είπε ο Μίτσελ, ο οποίος έθιξε τα ουσιώδα ζητήματα. Συμπληρώνω όμως ότι ασφαλώς ε, ο στόχος της προτάσεως προστηρίζεται από, το, από ένα πολύ ευρύ ε, φάσμα Βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε τις επιταγές του κανονισμού Μίμφιτ και έχουμε να εξετάσουμε ε, διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν πάντα με ομοιόμορφο τρόπο. Η Μαρίσα δεν είναι σκιώδης εντωμεταξύ βέβαια, είναι ε, έχει τη σύνταξη της νομοδότησης για την Ήτρε και φαντάζομαι ότι με διαφορετικό τρόπο θα χειριστεί τα θέματα των πρώτων υλών στην ενέργεια και το καθεξής. Εδώ έχουμε στο παράρτημα 3 ενσωματώσει όλα τα ζητήματα, αλλά δεν είναι σωστή η θέση αυτή για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων. Γι' αυτό προς την εισηγήτρια θα ήθελα να διατυπώσω το ερώτημα εάν θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το θέμα τη ΣΥΤΡΕ ως με, ρόλο γνωμοδότη, δηλαδή Επιτροπής Αρμόδιας για Γνωμοδότηση, θα πρέπει να το αναλάβουμε αυτοτελώς το ζήτημα αυτό. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, συνθήκες της διαμόρφωσης αγοράς και τον κίνδυνο της, ε, να παραλαπτεί η διαφάνεια. η συλλογή δεδομένων από αρχές οι οποίες μπορεί στη συνέχεια για να τις διαθέσουν, για να διαθέσουν τα στοιχεία αυτά, να ζητούν ένα τέλος, είναι κάτι το οποίο πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε. Το πώς δηλαδή αυτές οι αρχές θα μπορούν να ε, ελέγχουν τα στοιχεία, γιατί και στη διεθνή αγορά των πρώτων υλών δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε σωστά δείκτες αναφοράς και την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά. Δεν μπορεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπαγορεύει κανόνε για την Ασία ή τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Ρωσία και όλα τα κράτη του ΟΠΕΚ που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για τα οποία δεν βλέπω καμιά πιθανότητα να μα δίνουν στοιχεία ε, επακριβή. Εκτό και αν υπάρχει, εάν διαπιστώσουν ότι είναι λογική η νομοθεσία. Ε, άρα λοιπόν η διαφάνεια η οποία εχθές είδαμε ότι επευλήθησαν τα σχετικά ε, πρόστιμα, δεν είχαν... Ε, ε λοιπόν, οι όροι της διαφάνειας δεν είχαν τηρηθεί, γι' αυτό και επιβλήθη το πιο υψηλό πρόστιμο στην ιστορία 1,7 δις ευρώ. Άρα ναι, πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια για καλούς δείκτες αναφοράς, αλλά ταυτόχρονα πρέπει τα προϊόντα τα οποία συνδέονται με αυτούς τους δείκτες αναφοράς, επί παραδείγματι επενδυτικά κεφάλαια, παράκογα κτλ. να τα διαχωρίσουμε από τα υλικά αγαθά, όπως το πετρέλαιο και το καθεξής. Τα άλλα δηλαδή πρέπει να τα ξεχωρίσουμε από τα υλικά, γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες και σε αυτό ίσως χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση ο κανονισμός και θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε τι, ε, από τα παραρτήματα ποιο κομμάτι μπορεί να μπει μέσα στον κανονισμό, ποιο μπορεί να μείνει σε παράρτημα και πάνω απ' όλα τι μπορεί ε, στην πορεία της λειτουργίας του κανονισμού να τροποποιείται ως παράρτημα. Και πάνω απ' όλα, όπως είπα, ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή για τις πρώτες ύλες της ενέργειας. Κύριο Σμίτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την εξαιρετική αυτή έκθεση, όπως πάντα. Τώρα μιλάω από μια χώρα με μικρό νόμισμα μικρή χώρα με μικρό νόμισμα που έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία βέβαια γνωρίζετε και ορισμένες από τις τροπολογίες το φροντίζουν αυτό. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να το τονίσουμε και δεν άκουσα τον δανό μου συνάδελφο να το κάνει αυτό, οπότε το κάνω εγώ και για την Νορβηγία και για τον Κάιμπορ και για τον Νάιμπορ. Ξέρετε ότι αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να είμαι μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά δεν είμαστε στην Ευρωζώνη και η Λύρα είναι πολύ μεγάλο νόμισμα, αλλά η Σουηδική κορώνα όχι. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια κάποια νομοθεσία. Και βέβαια χρειαζόμαστε και αναλογικότητα και ευελιξία. Αλλά βλέπω πως ε, η τροπολογία σας αυτό το καλύπτει εν μέρη, αλλά θέλω να τονίσω για όλους. Τώρα δεν ξέρω την λεπτομέρειε λεπτομέρειες, αλλά για το Στάιμπορ στη Στοκχόλμη δεν υπήρξαν προβλήματα και λειτουργήσε. Εντάξει, Βέρνερ. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό που είπε και ο Γκέι Μίτσελ για τους πληροφοριοδότες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. και είδα ότι συμφωνείς και εσύ, Σάρον. Και φυσικά για τη διαφάνεια. Και είναι διασκεδαστικό να σας ακούει κανείς, γιατί όλοι μιλάνε για τη διαφάνεια. Έχει γίνει καραμέλα. Όταν εγώ πρώτα έγινα Ευρωβουλευτής το 1999, δεν ακουγόταν αυτή η λέξη. Η διαφάνεια μπορεί πάντοτε να προκαλέσει προβλήματα, όπως ξέρουμε. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά αυτούς που λένε πω, όποτε τι είπα. Πάντως σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ε, δημοσιονομικό, η διαφάνεια είναι ζωτική σημασία. Μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να υπάρξει κατάχρηση, αλλά αυτό συμβαίνει σπανίως μπορεί να πει ότι πρέπει να προσέχουμε, πάντως εν γέννη, η διαφάνεια είναι κάτι το πολύ καλό. Ευχαριστώ λοιπόν Σάρον. Ξέρω πως ε, επισκεφτήκε στο Στοκχόλμη, την Κοπεχάκη και το Όσλο. Βέρνερ. Μια και έκανε αυτή την ε, προσωπική αναφορά ο αγαπητός και αξιότιμος συνάδελφος Όλη Σμιτ ότι ήταν φιλελεύθερος ο Επίτροπος Μαγκρίβι, ο οποίος στην αρχή της ε, κρίσης αυτής της μεγάλης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής αντιδρούσε στην διαφάνεια. Και εμείς με το Κοινοβούλιο και την Περβός Περές συγκεκριμένα ζητούσαμε να έχουμε πολύ πιο καλές συνθήκες διαφάνειας. Μακάρι να μας είχαν ακούσει νωρίτερα. Αγαπητέ όλοι. Κύριο Σμιτ. Αγαπητέ συνάδελφοι. Τότε θα ήθελα και εγώ να απαντήσω ότι εμεί έχουμε στην Ιρλανδία και την Σουηδία διαφορετικές παραδόσεις, μάλλον από την Ιρλανδία στη Σουηδία υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Εμείς τη διαφάνεια την εισεγάγαμε στη Σουηδία το 1766. Να και ακούστηκε το όνομα της Ιρλανδίας, λέει ο κύριος Μέτσελ. Ότι όλοι αυτοί ήταν στη χώρα μου και μας τα είχαν κάνει μαντάρα πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω, να προσπαθήσω να απαντήσω. Καλωσορίζω και τις ε, τροπολογίες. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Ε, γιατί και όπως είπε και η Μίτσολ έπρεπε να δουλέψω γρήγορα σε αυτό το θέμα και είναι δύσκολο κανείς να με βρει γιατί συνήθως σε κάτι προεδρεύω, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω άλλες συνεδριάσεις ε, ταυτόχρονα και γι' αυτό και θέλω να έχω μια πολύ ευρία προσέγγιση για τις τροπολογίες και είπα ότι ε, θέλω να προσελκύσω τις απαντήσεις γιατί όλοι σκέφτονται πώς θα το αντιμετωπίσουν και όταν είπαν ε, ότι είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και γι' αυτό και έπρεπε να βγάλω και κάποια πράγματα όπως το κατόφλι για τα 100 δις ε, το... συμφωνώ μαζί σου Γκέι ότι ίσως πρέπει να δούμε ε, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησα να μείνω μακριά, να δούμε τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς και μετά να κάνουμε ένα είδος κατεξοδότηση πράξης για τα υπόλοιπα. Ε, αλλά μετά θεώρησα ότι δεν θα ήταν αρκετά ουσιαστικό αυτό. Θέλουμε πιο ουσιαστικό πλαίσιο. Αλλά δεν... Και θεώρησα ότι αυτό δεν θα σας ικανοποιούσε. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα του phasing των διαφόρων σταδίων που είχα και μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα τροποποιήσουμε κάποιες, κάποια, κάπως τη φύση των κατηγοριών και των νούμερων ώστε να είναι ας πούμε, αυτά απλά παραδείγματα και να φτάσουμε κάπως ε, πιο ε, σε κάπως πιο συγκεκριμένα πράγματα αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και κατευθύνες γραμμές για το πόσο τα κάνει όλα αυτά η ΑΚΑ. Ωστόσο για τους κρίσιμους δείκτες και για το ΚΑΙΜΠΟΡ, το ΚΑΙΜΠΟΡ δείχνει μάλλον ότι μπορεί να χρειαστεί να δούμε αν χρειαζόμαστε κάποιες φορές την αναλογικότητα ακόμα και εκεί. Και επίσης καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβουν αν είναι μέσα ή έξω, όταν είναι το, το κατόφλι, όταν δεν είναι τόσο ενεργό το κατόφλι. Τώρα, όσον αφορά στατιστικές υπηρεσίες και άλλα, εγώ είμαι της άποψης πως δεν πρέπει να τοποθετήσουμε εξαιρέξεις σοβαρές στην πρώτο επίπεδο, ούτε για τις κεντρικές τράπεζες και γι' αυτό τις έχω αφαιρέσει, αλλά θα ήθελα η να έρθει και να πει ναι, οι κεντρικές τράπεζες, οι κεντρικές στατιστικές υπηρεσίες έχουν τις δικές τους μεθόδους διακυβέρνησης και οι διατάξεις αυτές είναι αντίστοιχες και άρα λοιπόν γι' αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Θέλω να έχω κάποια σημεία, κάποια στοιχεία για να δούμε σε τι αντιστοιχούν αυτές οι διατάξεις. Ανησυχώ λιγότερο για τις στατιστικές υπηρεσίες, γιατί εκεί δημοσιεύονται τα πάντα όσον αφορά τους ελέγχους τον, ε, και τις διακυβέρνησης και τα λοιπά. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τις κεντρικές τράπεζες και θέλω τα δύο αυτά να ε, τα χειριστώ παρόμοια ώστε να έχουμε λίγο παραπάνω διαφάνεια για τις τράπεζες. Δηλαδή ποιες ακριβώς είναι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης, που λένε ότι είναι σωστό να βγεις από εδώ. Και το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει για άλλους. Έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ελαφρύ καθεστώς, επειδή υπάρχει ήδη άλλου είδους διακυβέρνηση ή ε, γιατί είναι προβληματικό για τον κώδικα διοντολογίας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ δύσκολο στην πράξη. Και πρέπει να έχουμε υπόψη τα διάφορα είδη δικτών αναφοράς που υπάρχουν. Έχουμε σχετικά λίγους συνεισφέροντας για κάποιους. Και εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να... και θέλουμε να ξέρουμε πάντοτε περισσότερα από το... για το τι συμβαίνει. Όταν έχουμε όμως χιλιάδες συνεισφέροντες, ε, πρόκειται απλά για στοιχεία που συλλέγονται και είναι δύσκολο να τα χειριστεί κανείς. Ξέρουμε ότι ε, έχουν γίνει απόπειρε και ότι έχουν αποτύχει, επειδή ακριβώς είναι τόσο πολλοί οι συνεισφέροντες και το κάνουν αυτό ε, θελοντικά. Αν λοιπόν κάτι δεν τους ενδιαφέρει απόλυτα μπορεί να μην συμμετέχουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να το ε, προχωρήσουμε σωστά. Τώρα για τους διαχειριστές. Θα πρέπει να γνωρίζεις ποιοι είναι οι συνεισφέροντές σου, διότι ε, πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, τίμοι, ε, επιχειρηματίες. Δεν είναι ο πάσα ένας που ξαφνικά θέλει να δώσει κάποια στοιχεία, οι διαχειριστές των δικτών φέρουν μια ευθύνη. Πρέπει να γνωρίζουν το κλάδο τους και να γνωρίζουν και την, τους συνεισφέροντες. Έτσι ώστε να είναι αντίστοιχο με τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένα οι δείκτες αναφορές. Επίση θα πρέπει να βλέπουμε ποιε είναι οι συνεισφορέ όταν ε, θεσπίζεται κάποια μεθοδολογία, όπω α πούμε για τι ανταλλαγέ. Υπάρχει ένα είδο κατεργασία από την ημερομηνία τη συναλλαγή και δεν υπάρχει τρόπο να επιβαρυνθούν υπερβολικά αυτά τα θέματα από τη στιγμή που έχουν αυτοματοποιηθεί, από τη στιγμή δηλαδή που έχει θεσπιστεί μια εποπτεία για τη μεθοδολογία. Πρέπει να γίνει δηλαδή εδώ περισσότερη δουλειά. Τώρα, για τα αγαθά είναι πολύ δύσκολο και πάλι και εδώ χρειάζεται ε, σταδιακή ε, εφαρμογή. Αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εδώ κάτι, εκεί όπου δηλαδή υπάρχουν ανησυχία, να χρησιμοποιήσουμε το, της της τη σταδιακή συμμόρφωση ώστε να μπορέσουν οι δείκτες να αναπτυχθούν όσον αφορά τα αγαθά και να συμμορφωθούμε με την ΙΟΣΚΟ. Προσπάθησα αυτά να τα τροποποιήσω με τον ίδιο τρόπο και στο παράρτημα 3. Αλλά πιστεύω πως αυτοί που εργάζονται από αυτόν θα μας δώσουν και περισσότερες ιδέες, γιατί ε, λόγω της ταχύτητας με την οποία χρειάστηκε να εργαστώ, εκεί πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν ε, το εξέτασα πολύ εις βάθος. Τώρα, για τους πληροφοριδότες, άρθρο 11 και ένα από τα παρατήματα, αν θυμάμαι καλά. και κώδικας διοντολογίας μαζί. Δεν έχω πρόβλημα με το να ενδυναμώσουμε αυτές τις διατάξεις και αν οι συνάδελφοι θέλουν να το κάνουν, συμφωνώ. Τώρα τα διάφορα συλλογικά σώματα. Προσπάθησα να το απλοποιήσω γιατί φοβούμαι πως μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη επιπλοκή των όσων συμβαίνουν και αν γίνονται πάρα πολλά μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω πως ε, τώρα απάντησα στα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε για το ρόλο της ΕΑΚΑ και πού και πότε αυτός μπορεί να ενισχυθεί, προσπάθησα να το σκεφτώ και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί η ΑΚΑ είναι πολύ μικρή και, και εύκολα μπορεί να τους επιβαρύνουμε υπερβολικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δημοσιονομικός ελεγκτικός ε, οργανισμός ε, που είναι μεγαλύτερος, στην ουσία θα το έβαζε στα πόδια αν έβλεπε ένα τέτοιο νομοθέτημα που έπρεπε να εφαρμόσει. Γι' αυτό και πρέπει εδώ και να κινηθούμε προσεκτικά. Εγώ θα έλεγα δεν έχω πρόβλημα η ΑΚΑ να βγάζει τις κατευθύνες γραμμές και να ορίζει προς τα που θα κινηθούν και οι ελληνικές αρχές. Ίσως να υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι χώροι όπου σημαντικοί δείκτες αναφορές που είναι διασυνοριακοί με την έννοια από πού συλλέγονται οι πληροφορίες, από πού προέρχονται οι πληροφορίες, αλλά και πάλι μπορεί και αυτό να φανεί ότι είναι υπερβολικά μεγάλο έργο για την ΕΣΜΑ η ΕΑΚΑ. Είναι όπως ο μηχανισμός της σταθερότητας κάπως, όπου η ΕΚΤ έχει τη γενική ευθύνη, αλλά για κάποια πράγματα τα αναθέτει στα κράτη-μέλη και πάλι. Αν θέλετε, εδώ ανατίθονται περισσότερα πράγματα αλλά ίσω αυτό δεν είναι ο τρόπο για να προχωρήσουμε, ίσως αυτό να λειτουργήσει καλύτερα. Και έχω και μια σχετική διάταξη, ότι αν αρμόδια αρχή θεωρήσει πω μπορεί κάτι να γίνει καλύτερα από την ΕΣΜΑ, να έχει τη δυνατότητα η ΕΣΜΑ να το κάνει. Να δούμε λοιπόν τι προτάσει θα κάνουν και οι συνάδελφοι για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πάντω είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Αν τα αφαιρέσουμε όλα από την ΕΑΚΑ, ε, θα έχουμε ε, σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομεί. Θα δούμε ενδιαφέρον ε, τι θα γίνει στην Ήτρε. Για, λόγω των αγαθών έχουμε προβλήματα όπου τα πράγματα είναι απλά τιμές και μετά ξαφνικά γίνονται δείκτες. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Το γνωρίζω πολύ καλά και όσοι έχετε κάνει τη σχετική εργασία σας είμαι ευγνώμων. Νομίζω πως αναφέρατε επίσης αυτή την ε, μείωση των ε, συνεισφορών. Αν λες στον ε, συνεισφέροντα ότι υπογράψτε στη, εδώ σε αυτή τη σειρά και μετά είστε νομικά υπεύθυνοι, φαντάζομαι ότι θα εξαφανιστούν και άρα δεν θα έχουμε τη συνέχεια που χρειαζόμαστε. Επίσης αναρωτήθηκα αν υπάρχει μεγαλύτερη ε, σχέση, κάτι που πρέπει να κάνουμε στους ορισμούς για το ποιοι θα εποπτεύονται, ποιες οντότητες θα εποπτεύονται και ίσως να έχουμε και εκεί κάποιες κατηγορίες με συγκεκριμένες εντολές. Οπότε αρχίζουν όλα κάπως να γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που στην Επιτροπή Βιομηχανής μπορεί εδώ να με βοηθήσουν με κάποιες τροπολογίες και ο Βέρνερ ανέφερε, το θέμα της πώληση στοιχείων που κάλυψα. Δεν μπορούμε να, να μειγνύουμε πυρογγελματικά ε, Θεμητέ ε, επαγγελματικέ ε, προστασίες. Θα έχουμε κάπως στεναρή άποψη όσον αφορά την ε, πνευματική ιδιοκτησία και πολλές φορές αυτή επεκτείνεται και σε πράγματα που δεν θα έπρεπε, αλλά θα το εξετάσω πολύ σοβαρά γιατί εδώ υπάρχει γνήσια ανησυχία. Δεν ζήτησα στην Κομισιό να παρέμβει γιατί έχουμε κάπως καθυστερήσει. Πάντως αν οπωσδήποτε θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να το κάνει συντόμως και όποιες ιδέες προέλθουν από την Κομισιόν για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από τα προβλήματα που ανέφερα και που ανέφεραν και οι συνάδελφοι θα το δούμε με ενδιαφέρον γιατί όπως είπα όσο πιο πολλές πληροφορίες έχουμε τόσο καλύτερα. Πιθανότατα θα πρέπει να κάτσω την Κυριακή να τα δω όλα αυτά για να σκεφτώ πώς θα ταιριάξουν όλες αυτές οι τροπολογίες όσοι ακούν, παρακαλώ να μου δώσουν τις πληροφορίες που θέλουν γρήγορα γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο. Η προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι 5 το απόγευμα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα τη συζητήσουμε στις 20 Ιανουαρίου με στόχο να ψηφίσουμε στις 30. Αυτό σημαίνει πως αν το Συμβούλιο θελήσει να κοιτάξει αυτό που κάναμε και να μας πει τη γνώμη του, θα μπορούσαμε γρήγορα να τελειώσουμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Διαφορετικά θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και βεβαίως τότε θα είμαστε έτοιμοι για να αναλάβει το θέμα το επόμενο Κοινοβούλιο να καλέσω ίσως την Προεδρία, επειδή προς, κινούμεθα προς μια συνενετική λύση, να εξετάζει τις ε, ιδέες μας και να αρχίσουν να το σκέφτονται τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι και τώρα περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, το κοινό σύστημα φόρο προστιθέμενης αξίας. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης του Ιβο Στρέιτσεκ. Ας περιμένουμε να φύγουν όσοι θέλουν για να μπορούμε να μιλήσουμε με ησυχία και να μην χρειάζεται να φωνάζει ο Ήβο. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind and nice of you. Ό,τι ευγενικοί που είστε. Φεύγετε με μεγάλη ησυχία. Ο Ήβο για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. No, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, ρίχνοντας μια ματιά γύρω μου βλέπω ότι έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος. Καλό σημάδι αυτό. Αυτό δείχνει ότι η έκθεση δεν είναι επίμαχη. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Και θα είναι θερμή υποστήριξη των Ευρωβουλευτών από όλε τι πολιτικές ομάδες για την έκθεσή μου. Ο φόρος προστιθέμενης αξία είναι σχετικά πρόσφατο φόρος στην ιστορία των φόρων. Ένα φόρος όμως ιδιαίτερα προσφυλής στους Υπουργού Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι αντίθετα δεν πεθαίνουν και όλα για το ΦΠΑ, ενώ οι διοικήσει ε, βλέπουν και υπέρ και κατά. Ο φόρος προστιθέμενης αξία εξασφαλίζει κάποια έσοδα στο κράτος, αλλά υπάρχουν ε, πολλές ε, δυνατότητες απάτης και κατάχρησης του φόρου. Άλλο αρνητικό σημείο είναι η περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις για το ΦΠΑ. και είναι εύκολο κανείς δεδομένης αυτής της περιπλοκότητας να αποφύγει τις φορολογικές του ευθύνε. Πάντως η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ αξιόλογη. Καταρχήν ε, είναι ευανάγνωστη, εύληπτη και καθόλου αφιλεγόμενη. Πολύ καλό λοιπόν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεωρώ ότι θα είναι και πολύ εύχριστη αυτή η πρόταση και θα βοηθήσει τα μάλλα στις ε, διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Μερικές φορές βέβαια είναι δύσκολη η δήλωση και η καταβολή και η απόδοση ΦΠΑ όταν μιλούμε για διασυνοριακές συναλλαγές. Γι' αυτό καλό θα είναι να εξασφαλιστεί μια ομοιομορφία στις δηλώσεις. Έχουμε βασικές αρχές που καλό θα τα ανατηρηθούν. Μία απλούστευση, για παράδειγμα, των διαδικασιών. Μάλιστα, χάρη στον ηλεκτρονικό μορφότυπο και στην τυποποιημένη δήλωση θα εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια. Και για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ είναι μια εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. Είτε αυτό αφορά αγαθά είτε υπηρεσίες. Επίσης ε, και οι εθνικές εφορίες θα μπορούν να εισπράττουν ευκολότερα το ΦΠΑ. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση που θα διευκολύνει τους επιχειρηματίες αλλά και τις διοικήσεις. Αν έχετε κάποια εμπειρία από διασυνοριακό εμπόριο θα γνωρίζετε ότι Πολύ συχνά είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις φορολογικές νομοθεσίες ε, των χώρων μελών. Μία άλλη χαρμόσυνη είδηση για τα Υπουργεία Οικονομικών είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα οδηγήσει εξοικονόμηση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τις διοικητικές δαπάνες επεξεργασίας των δηλώσεων. Διόλου αμεληταία λοιπόν αυτή η οικονομία και πολύ ευχάριστη είδηση για τα Υπουργεία Οικονομικών. Εδώ προτείνουμε ένα ελάχιστο όριστο υποχρεώσεων με πέντε στήλες για συμπλήρωση σε αυτή την τυποποιημένη δήλωση. Ένα έντυπο που είναι σίγουρα απλούστερο και ευκολότερο για τις επιχειρήσεις ε, που χρειάζεται να τηρήσουν διάφορες φορολογικές παραδόσεις. Προβλέπεται ένα ελάχιστο αριθμό πληροφοριών που απαιτούνται σε αυτή τη δήλωση, την τυποποιημένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ε, διαφορές ε, και τις ιδιαιτερότητες της φορολογικές παραδόσης των κρατών μελών και κατέληξε σε μια πολύ ελαστική πρόταση. Έτσι, μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες όταν αυτό απαιτείται, αλλά και αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες ε, θα υποβάλλονται με βάση ενιαίο μορφότυπο με βάση τυποποιημένη, τυποποιημένη δήλωση. Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, προβλέπεται ένας μήνας για την υποβολή της δήλωσης και η πρόταση λαμβάνει υπόψη ότι για τις μικρές επιχειρήσεις μπορεί να παραταθεί η προθεσμία. Να αφήσουμε ένα τρίμηνο στις μικρές επιχειρήσεις για να υποβάλουν τη δήλωση ΦΠΑ, για να μην τις επιβαρύνουμε υπερβολικά. Εν κατακλείδη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ αξιόλογη, εύχριστη, πρακτική, μειώνει τη γραφειοκρατία, εξασφαλίζει μεγάλες οικονομίες, περιορίζει τις διοικητικές δαπάνες Και το βασικό είναι ότι περιορίζει και τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Ιδιαίτερα σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, κάτι που είναι πολύ θετικό. Και ε, ευχαριστώ εκ των προτέρων τους σκιώδης ηγητές για τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της έκθεσης. Ευχαριστώ θερμά και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ εξόλογο υλικό που μας μοίρασε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Γεια Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ΕΣΑΙΑ μου ζήτησε να διατυπώσω τις δικές της προτάσεις και θέσεις για να καταγραφούν στα πρακτικά. Ε, θεωρεί λοιπόν ότι είναι ευπρόσδεκτες ε, και την κατάλληλη στιγμή προτάσει Επιτροπής, αποδεκτή η πρόταση του συγητή, αν και οι τοποθετήσεις για το Ταμείο Καρουσέλ ίσως χρειάζονται πιο πολλές διευκρινήσεις. Επίσης μας λέει ότι χρειάζεται να είναι καλή διατύπωση των προτάσεων της Επιτροπής. Έχει κάποια σχόλια μόνο, τα οποία είναι τα εξή. Με βάση τις προτάσεις θα πρέπει πέντε ε, πληροφορίες να προσφέρονται σε κάθε δήλωση ΦΠΑ υποχρεωτικά και μπορούν τα κρατη να συμπληρώσουν άλλα οκτώ πεδία πληροφοριών ε, ανάλογα με τις ε, προτάσεις τους. Συνολικά λοιπόν 13 πεδία πληροφοριών για τις δηλώσεις ΦΠΑ που όμως έτσι δεν θα είναι ε, ισοδύναμες για κάθε κράτος μέλος, μόνο στις 5, στα 5 υποχρεωτικά πεδία πληροφοριών. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί επιπλέον ε, τι είδους απαιτήσει έχει το κάθε κράτος μέλος από τις επιχειρήσεις και άρα δεν θα είναι ισοδύναμο το πεδίο. Και αυτό προτείνει η κυρία Σάγια να περιοριστεί ακόμη περισσότερο το πεδίο, ο αριθμός αυτών των πεδίων πληροφοριών κατά την επεξεργασία της προτάσεως Επιτροπής. Έχουν διαφορετικούς κανόνες για το ΦΠΑ τα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να προσφέρουν σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για το τι πρέπει να καταγράφεται σε κάθε πεδίο του κανονισμού ΦΠΑ. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, κατά προτίμηση όμως σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζουμε, Πρόεδρε, ότι όταν ε, ξεκινήσει το έργο για, το, ε, για τη διαδικτυακή πύλη του ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα, επιληθούν, θα έχουν επιληθεί αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτό το βλέπουμε να σημαίνει πολύ σύντομα. Επίση, θα πρέπει οι επιχειρήσει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος και αυτές βέβαια οι ηλεκτρονικές δηλώσεις ΦΠΑ θα πρέπει να ενταχθούν για το κάθε κράτος ε, σε ένα αποδεκτό σύστημα ηλεκτρονικής ε, υπογραφής και βέβαια η ηλεκτρονική αρχιοθέτηση θα πρέπει να προχωρήσει. Αν και όπως λέει η κυρία Σάια δεν είναι βέβαιο το πώς θα μπορέσουν να χειριστούν όλο αυτό τον αυτοματισμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά βέβαια ο αυτοματισμός όπως και να είναι είναι κάτι θετικό για την κυρία Σάια προσβλέπει σε μια καλή και επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή, ο οποίος έχει από ό,τι βλέπει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο έργο αυτό και πιστεύει ότι μπορεί να καταλήξει συμφωνία χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο το λόγο. Η Επιτροπή μου πώς να τοποθετηθεί. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστώ τον κύριο, ευχαριστώ τον κύριο Στράτσο και το εξαίρετο το έγγραφο και την υποστήριξη στην πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι είναι ένα μέτρο σημαντικό. Ε, βλέπουμε ότι μπορεί δηλαδή να σημάνει κέρδος έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από ε, διοικητική επιβάρυνση κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν τις πιο μικρές από αυτές. Ε, πρόκειται για μια πρόταση η οποία μπορεί να διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο ιδιαίτερα και να συμβάλλει στον περιορισμό της, ε, του, ε, της απόκλησης μεταξύ του θεωρητικού ΦΠΑ και των πραγματικών εσόδων ΦΠΑ και αυτό δεν αφορά μόνο τις απάτες αλλά γενικά τα προβλήματα έχουμε να κάνουμε 193 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση πρόσφατη μελέτη δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Θέλετε να λάβετε το λόγο πάλι. Ε, Μια-δύο προτάσει αν μου επιτρέπετε. Και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με τους ε, λοιπούς και Και στα όσα ανέφερε ο Γκέι, είναι εύκολο να λυθούν ε, οι επιφυλάξεις της κυρίας Σαϊά δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαι απολύτω σίγουρος ότι θα βρούμε λύσεις. Καλώς, ευχαριστώ. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. 5 το απόγευμα, 16 Δεκεμβρίου. Συζητούμε στις 22 Ιανουαρίου. Ψηφίζουμε στις 3 και δεύτερη ολομέλεια Φεβρουαρίου με βάση το ισχυρό χρονοδιάγραμμα. Αλλά έχουμε τώρα τον κύριο να κανονικά στο πρόγραμμα με τον διάλογο ε, για τις 11.30 προβλέπουμε. Επομένως διακόπτω και παρακαλώ και εσείς αλλά και άλλοι να είστε στην αίθουσα εκείνη την ώρα για τη συζήτηση μαζί του.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 Σε Okay. Um, if we, if we, shh, shh, shh, shh. Um, we're, we're also happy to see our, our, our... Με χαρά βλέπουμε και τον πρώην αντιπρόεδρο εδώ και τον καλούμε να καθίσει στη θέση του. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε πανευτυχείς ε, που έχουμε πάλι κοντά μας τον Έντουαρτ στην Επιτροπή μας. Σχεδόν κάθεται στην ίδια θέση. Εδώ καθόταν και ως αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ. Και τον ευχαριστώ θερμά και για το έργο που είχε επιτελέσει τότε, ιδιαίτερα στα θέματα της στατιστικής. Τώρα έχει προχωρήσει σε άλλα θέματα. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Και μια και είναι πέμπτη και πολλοί συνάδελφοι χρειάστηκε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είμαστε και πιο χαλαροί. Είμαστε λιγότεροι, πιο χαλαροί. Θα ακούσουμε λοιπόν τα εισαγωγικά σας σχόλια και μετά θα έχουμε γύρους ερωταπαντήσεων. Έτσι θα έχεις χρόνο να πτύξεις κάποια σημεία και αργότερα και στο τέλος σε ακούμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα πάντως που ήρθες. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Σάρον και εγώ αισθάνομαι πανευτυχής που επιστρέφω στην ΕΚΟΝ. Εθήτευσα τέσσερα χρόνια κοντά σας. Τώρα είμαι σε μια θέση που υποτίθεται ότι πρέπει να εφαρμόσω αυτά που λέγαμε στην Επιτροπή. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γεια σου Λίζα, Ελίζα. Δηλαδή χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση, ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέτρα που θα ενισχύουν, θα τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη αποφυγή του διλήμματος λιτότητας ε, απέναντι στην ανάπτυξη. Αρχίζουμε και εφαρμόζουμε αυτό που συζητούσαμε επί εβδομάδες ολόκληρες, το δίπτυχο πακέτο. Τώρα είμαι από την άλλη πλευρά του τραπεζιού και καλούμε να το εφαρμόσω. Και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την ανταλλαγή απόψε μαζί σα. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τη διαδικασία του υπερβολικού χρέου Και η πατρίδα μου κάνει μια δειγματοληψία από όλα αυτά τα θέματα. Το τελευταίο 9 πάσαμε και ένα ρεκόρ, γιατί ξέρω ελάχιστους υπουργούς οικονομικών που χρειάστηκε να υποβάλουν και να εγκρίνουν δύο προϋπολογισμούς μέσα στον ίδιο χρόνο. Γιατί ο πρώτος απορρίφθηκε, ο πρώτος που υποβάλαμε το Μάρτιο. Χρειάστηκε να τον αναθεωρήσουμε, να τον επανυποβάλουμε, να τον επαναφέρουμε στην πραγματικότητα για να περιλαμβάνει και ρεαλιστικές προγνώσεις ε, για την οικονομική ανάπτυξη, για τα έσοδα, για το έλλειμμα. Όλα αυτά τα θέματα έπρεπε να αναθεωρηθούν στον διορθωμένο προϋπολογισμό. Πολλό δε μάλλον που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Ε, το ότι η Μάλτα δηλαδή για μία ακόμη φορά περιέπεσε σε υπερβολικό χρέος, στην παγίδα του υπερβολικού χρέους και άρα θα πρέπει να υπαχθεί στη διαδικασία του υπερβολικού χρέους. Μετά από μήνε βέβαια μα ανήγγειλε ότι κατάφερε να αναρρώσει, να ξεφύγει από αυτό. Πολύ ενθαρρυντικό για την Επιτροπή. Μάλλον μα έφερε σε δύσκολη θέση γιατί έχουμε και τι προεκλογικέ εκστρατείε, την πολιτική αστάθεια. Ιδιαίτερα όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ε, πολύ ασθενής, με οριακή πλειοψηφία έπεσε η κατανάλωση, μειώθηκαν ε, τα εισοδήματα, ενώ οι δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες. Οπότε οι προβλέψεις ε, για 2,5% μετατράπηκαν σε 3,3% του ΑΕΠ. Τότε η οικονομία φαίνεται ότι προχωρούσε. Αργά, αλλά σταθερά και μάλιστα όταν μίλησα με τον Όρι Ρεν, το παρομοίωσε, την οικονομία με ένα πλοίο ιστιοφόρο που έπρεπε να κινηθεί με πολύ ασθενή άνεμο. Αλλά έστω και τη λίγη αυτή όθηση έπρεπε να την αξιοποιήσουμε, ήταν πολύ σημαντικό. Συναντήθηκα με τον Όλι Ρεν και εξετάσαμε την πιθανότητα να υποβάλουμε προϋπολογισμό με δρακόντιες περικοπές και είπαμε ότι θα λάβουμε πολύ αποτελεσματικές δράσεις και θέλαμε μέχρι το 2013 να έχουμε περιορίσει το έλλειμμα κάτω από 3, το χρέος κάτω από 3%. Δεν ήταν και πολύ αξιόπιστο αυτό για την Επιτροπή, γιατί οι δικέ σου προβλέψει ήταν 3,4 για φέτο, 3,5 για το χρόνο, αλλά εμείς κάναμε σωστά τους υπολογισμούς μας πήραμε τα μέτρα μας και είπαμε ότι φέτος θα, τελειώσουμε το χρόνο με χρέος κάτω από 3% Και υποσχεθήκαμε ότι θα αναλάβουμε δράση, αλλά με το δικό μας τρόπο. Και αντί να περικόπτουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, κοινοφελείς υπηρεσίες ή να ενοχλήσουμε κάποιες ομάδες ή να αγγίξουμε λεπτές πολιτικές χορδές και να δημιουργήσουμε δυσπιστία, αποφασίσαμε να τονώσουμε την οικονομία, γιατί όταν αρχίσει να πέφτει το ΑΕΠ, τίποτα δεν μπορεί να διορθώσει, να αναχαιτήσει την, την κατρακύλα και να επιτρέψει την ανάκαμψη και την ισορροπία των ε, δημοσίων λογαριασμών. Και τελικά καταφέραμε και πείσαμε τον Όλυ Ρεν και όντως λάβαμε αποτελεσματικά μέτρα. γιατί τη 20 εκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε περικοπές και οικονομίες σε 20 εκατομμυρίων. Περιορίσαμε τις ε, σπατάλες τις υπεραισιόδοξες αιτήσει για χρηματοδότηση. Και δώσαμε λεπτομεριακή ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 1η Οκτωβρίου, όταν χρειάστηκε να υποβάλουμε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης και την έκθεση αποτελεσματικής δράσης, δύο εκθέσεις έπρεπε να υποβάλουμε για την 1η Οκτωβρίου, Περιγράψαμε με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τομείς στους οποίους κάναμε τις περικοπές και γιατί πιστεύουμε ότι θα τελειώσουμε το 2003 με χρέος κάτω του 3%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τις δικές της απόψεις και αντιδράσεις στην έκθεσή μας για την αποτελεσματική δράση και δήλωσε ότι όντως ήταν αποτελεσματικές οι δράσεις μας, οπότε δεν χρειάζονταν περαιτέρω διαβήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Μάλτας, για φέτος τουλάχιστον. Τώρα, τι θα γίνει του χρόνου είναι θέμα σχεδίου προϋπολογισμού. Αυτό το υποβάλαμε όπως και οι υπόλοιπε χώρες στα μέσα Οκτωβρίου και είπαμε ότι οι διαρθρωτικές μας προσπάθειες που μας ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το διπλό παχέτο, το 0,6 για την διαρθρωτική ισορροπία, ε, υποσχεθήκαμε ότι θα πέσουμε κάτω από το 3%, θα φτάσουμε στο 2,1% του χρόνου. Ποιοι ήταν οι στόχοι της κυβέρνησης τώρα. Η νέα κυβέρνηση έπρεπε να εξετάσει τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Μερικές φορές συμφωνούμε με αυτές τις συστάσεις, άλλες φορές διαφωνούμε. Στην περίπτωση τη δική μας θεωρήσαμε ότι οι συστάσεις ε, αντικατόπτρισαν μία αντικειμενική αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των εικοναξιολόγησης, αξιολόγησης, και πραγματικά περιοριζόταν στα ουσιώδη προβλήματα της Μάλτας. Το πρώτο, η πρώτη σύσταση αφορούσε τη δημοσιονομική διακυβέρνηση, φορολογική διακυβέρνηση. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στο τέλος. Βέβαια, οι ανάγκες της χώρας ε, ήταν πολλές. Η πρωταρχική είναι η ενέργεια η Μάλτα είναι νησί, εξαρτάται από το πετρέλαιο με πολύ ρευστέ ε, τιμές. Και επίσης ε, είχαμε πολύ αναποτελεσματικά εργοστάσια. Μερικά ήταν μόνο 30% από την ποσότητα που κανονικά έπρεπε να παράγουν. Επίσης δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Η, η κυβέρνηση σκέφτηκε να στραφεί και προς το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αγωγό με τη Σικελία. Αν και ελπίζουμε ότι σε 5-6 χρόνια θα συνδεθούμε με τη Σικελία με αγωγό φυσικού αερίου. Πάντω προ το παρόν και πιστεύουμε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα καταφέρουμε να έχουμε διαφοροποίηση και προ το φυσικό αέριο, ώστε να κάνουμε οικονομίε ε, της τάξης του 35%. 25% των οικονομιών θα μετακυληθεί στον κλάδο και στους καταναλωτές εν το χρόνο. Επίσης θα έχουμε ε, μία σύνδεση Σικελίας Μάλτας. Ε, οπότε θα έχουμε όχι μόνο πετρέλαιο, θα έχουμε και μία σύνδεση με τη Σικελία και το φυσικό αέριο. Έτσι θα βελτιωθεί το ενεργειακό τοπίο της Μάλτας, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Οπότε αντιμετωπίζουμε έτσι την δεύτερη σύσταση, την ειδική για τη Μάλτα, που ήταν πολύ σημαντική. Ένα συναφές θέμα αφορά την ενεργειακή παραγωγή που είχε σχεδόν χρεοκοπήσει. Δηλαδή δεν μπορούσε να αποπληρώσει ένα αναπτυξιακό δάνειο της Γερμανίας που είχε συναυθεί πριν 25 ετία και αν δεν το είχαμε σώσει θα είχε χρεοκοπήσει και θα είχε συμπαρασύρει στη χρεοκοπία ολόκληρη τη Μάλτα. Αναζητήσαμε ένα στρατηγικό εταίρο, τον βρήκαμε στο πρόσωπο των Κινέζων που εκδήλωσαν προθυμία να γίνουν ένα στρατηγική εταιρεία, αναλαμβάνοντας ε, ένα μερίδιο μειοψηφία μετοχικό. Βέβαια θα δούμε ποιο θα είναι αυτό το μερίδιο, δείχνοντας τη σωστή επιμέλεια. Πάντως η επιπτώσει όχι για τον παραγωγό ενέργεια, αλλά για την κυβέρνηση, η Μάλτα το 60% του ΑΕΠ το είχε σε παθητικό εκτάκτο ανάγκης και εξακολουθεί να το έχει contingency liability. Θέλουμε να το υποδιπλασιάσουμε, γιατί θα δοθούν 200 εκατομμύρια. Έχουμε ένα υψηλότερο χρέος, 850 εκατομμύρια από το 1 δισεκατομμύριο είναι το κόστος αυτού του, αυτού του ομίλου του ενεργειακού. Οπότε θα μειώσουμε τελικά το παθητικό εκτάκτο ανάγκης της χώρας σε αισθητά με την σύναψη αυτής της εταιρικής σχέσης και αυτό αναγνωρίστηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Δεύτερο σημείο. Αύξηση του δυναμικού της οικονομικής ανάπτυξης, γιατί έπεφτε το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης μάλιστα σταθερά. Από 4% το 2000 φτάσαμε στο 1,5%. Ο λόγος ε, της ύφεσης είναι ότι ε, στηρίζεται στο μισθολογικό κόστος σε επενδύσεις και την παραγωγικότητα. Αυτές είναι οι βασικές συνιστώσεις της οικονομικής ανάπτυξης της ε, Μάλτας. Ήταν σαφές όμως ότι η Μάλτα με, το, με τη χαμηλότερη συμμετοχή σε εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πρόβλημα. Και η ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό επίσης ήταν ε, σημαντικό πρόβλημα. Όλα αυτά θα ήλθαμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο νέο προπολογισμό έχουμε μια σειρά μέτρων που στόχο έχουν να ενισχύσουν το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, αλλά και γενικώ στην αύξηση του εργατικού δυναμικού. Μάλιστα θα ε, εισαγάγουμε δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς, δαπανηρό μέτρο, αλλά πολύ αποδοτικό κοινωνικά και θα έχει αντίκτυπο θετικό στην οικονομία. Επίσης, ε, θα, θα προβλέψουμε ε, βρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα για τη φροντίδα των παιδιών που θα λειτουργούν και το απόγευμα μετά τη λειτουργία δηλαδή, του σχολικού ωραρίου. Έτσι θα βοηθήσουμε μητέρες ή γονείς που θέλουν να εργαστούν να μην χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιος θα φροντίζει τα παιδιά. Και μάλιστα ε, παρατείναμε κατά δύο εβδομάδες την ε, άδεια μητρότητας. Αυτό έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση με την αμέριστη συμμετοχή και υποστήριξη και της ε, αντιπολίτευσης. Εμείς θεωρούσαμε ότι μία μικρή άδεια μητρότητας θα ενίσχυε την οικονομία. Επίσης, για τις γυναίκες άνω των 40 έχουμε κάποια φορολογικά κίνητρα και μία πολύ ε, ενεργό στρατηγική. Επίσης, ε, προσθέσαμε ένα άλλο σύστημα για την αξιοποίηση της εργασίας. Το θέμα όσων λαμβάνουν επιδόματα ε, είναι ότι δεν εργάζονται. Οι άνθρωποι όμως είναι λογικοί. Δεν είναι τεμπέληδες, είναι λογικοί. Δεν θέλουν να εργάζονται γιατί δεν τους εξυπηρετεί αυτό. Τώρα ε, αφαιρέσαμε τα επιδόματα για μία τριετία. Όσοι βρίσκουν δουλειά θα κρατήσουν ένα των επιδομάτων αυτών, αλλά με μία σταδιακή μείωση για μία τριετία. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η μεταφορά της φορολογίας από την εργασία στην κατανάλωση. Δηλαδή, μειώσαμε και θα συνεχίσουμε για μία τριετία τη, τη φορολογία των, μέσω, των εισοδηματιών της μέσω επίπεδου και σταδιακά αυξήσαμε τους φόρους της κατανάλωσης, ε, έμεσους φόρους κατανάλωσης ε, που αυξήθηκαν φέτος. Αυτό θα απαλλάξει την εργασία από το φορολογικό κόστος, ενώ θα αυξηθεί χάρη στους φόρους κατανάλωσης η οικονομική ανάδειξη, ό,τι αφορά την ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Η Μάλτα πάλι είναι ουραγός. Έχουμε τον υψηλότερο λόγο ε, εγκατάλειψης ε, των σπουδών. Έχουμε καλό πολυτεχνείο, καλό πανεπιστήμιο, αλλά παρόλα αυτά στο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές δεν φτάνουν μέχρι το απολυτήριο ηλικία, οπότε είναι άχρηστη για την αγορά εργασίας. Γιατί η αγορά εργασίας απαιτεί, αν μη τι άλλο, Στοιχείο ηλικίου, απολυτήριο ηλικίου. Οπότε, σε συνδυασμό με την εγγύηση των νέων, εφαρμόζουμε μια πιο ενεργό στρατηγική για να εμποδίσουμε την πρόορη κατάληψη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι έτσι θα ενισχύσουμε και την αγορά εργασίας. Τώρα, το επόμενο είναι αυτό που είναι το τι προσελκύει τι επενδύσει. Χρειάζεται μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη και εδώ πάλι η Μάλτα είχε τη μακρύτερη περίοδο ε, για υποθέσεις που ολοκληρώνονται, που εκδικάζονται και εδώ μόλις ολοκληρώθηκε η έκθεση σχετικά με την ε, μεταρρύθμιση τη ΤΑΡΑ ε, που ανέλαβε ένας εισαγγελέα και επίσης μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Ε, προσπαθούμε να δούμε τι αποτελεί εμπόδιο για μεγαλύτερε επενδύσεις στη Μάλτα Έχουμε επίσης εδώ μια κάποια συμφωνία γιατί είχαμε μια μεταρρύθμιση πριν από κάποια χρόνια και αυξήσαμε το συντάξιμο όριο στις, 65. Ε, Θέλουν κάποιοι να το αυξήσουν περισσότερο, πολιτικά όμως υπάρχει αντίσταση, αλλά μεταξύ τον επόμενο του χρόνου θα εισάγουμε το τρίτο της του πυλώνα στη Μάλτα που δεν υπήρχε παλιότερα. Έχουμε ολοκληρώσει την νομοθεσία και ε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Κλείνοντα και ίσω να απαντήσω και στις ερωτήσεις ε, τώρα για το υπερβολικό έλλειμμα και τη σχετική διαδικασία, γιατί αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Καταρχήν, ε, προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμφωνία με την Κομισιόν. Όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, όταν είμαστε εδώ, είμαστε αρκετά επικριτικοί κατά οποιοδήποτε ήταν εξαιρετικά ε, ε, αισιόδοξο για την ανάπτυξη, για τα έσοδα ε, σε σχέση με τα όσα σενετά προέβλεπε η Κομισιόν. Αυτή τη φορά το κάναμε ανάποδα. Η Κομισιόν προβλέπει υψηλότερη ανάπτυξη οικονομική από το Υπουργείο μας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα γιατί τουλάχιστον δεν προβλέπουμε υψηλότερα εισοδήματα και άρα οι δαπάνες είναι πιο ελεγμένες. Ε, έπειτα όμως έχουμε συμφωνήσει για ένα σφάλμα που πιστεύουμε ότι έκαναν για, τις, ε, για την φοροαποφυγή. Εμείς από το πλευρά του Υπουργείου ξέρουμε από το Ταμείο τι εισέρχεται και τι δαπανάμε και ξέρουμε ότι είμαστε εντάξει. Εμείς λέμε πως αφήστε να τελειώσει ο χρόνος και το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του. Και έπειτα, στην ερηνή πρόβλεψη ελπίζουμε πως αυτό θα αναθεωρηθεί με βάση την πραγματικότητα. Σε αυτά θα νομίζω θα σταματήσω. Έχω που και άλλα να πω αν θέλετε για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όντως είναι μεγάλη χαρά να ακούμε τις επιτυχίες σας, για τις επιτυχίες σας και βέβαια που βλέπετε τις δυσκολίες. Είναι λυπηρό βέβαια το ότι, όπως λέτε, αναζητήσατε εταίρους στην Κίνα. Ενώ το πρόβλημα ήταν η δυσκολία αποπληρωμής ε, δανείου προς Γερμανική τράπεζα. Θα ήταν καλύτερο να είχε μείνει εντός ε, του οίκου μας όλη αυτή η ιστορία, όπως λένε. Ε, θα γίνει συζήτηση τώρα με πρώτα τους συντονιστές, μετά θα έχουμε και τη διαδικασία καρστιά. Ζωμπόλ, θες να πάρεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όχι ερώτηση. Απλώς θέλω να καλωσορίσω εδώ τον παλιό φίλο που έγινε και υπουργό και να τον ευχαριστήσω για την πολύ σαφή παρουσίασή του, την ειλικρινή αυτή έκθεση της κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετώπισε η, Μάλκα, η Μάλτα και τον καλούμε βεβαίως να υλοποιήσει την στρατηγική και την πολιτική όπως την προβλέπει ο ίδιος με την ελπίδα ότι θα επιτύχει. Λίσσα. Όντως είναι χαρά που σας βλέπουμε εδώ σε αυτά τα νέα καθήκοντα, σε αυτή τη νέα θέση. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε την ανάλυση των πρακτικών ζητημάτων που σας απασχόλησαν. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που αναφέρατε και τα σχόλια της Πρόεδρου. Και εμείς στην Πορτογαλία έχουμε αντίστοιχη στρατηγική. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την συμμετοχή της πολιτείας στο, στην ενέργεια και τώρα έχουμε την συμμετοχή κινέζικων επιχειρήσεων. Αλλά μπορούμε τουλάχιστον να δούμε με τη στρατηγική ο ένας και ο άλλος τι είδους αποτελέσματα μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς όσο και σε εμάς βέβαια. Αναφέρεστε επίσης σε κάποια στοιχεία όπου συμφωνείτε και άλλα όπου διαφωνείτε με την Επιτροπή. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την ανάγκη να μην παρασυρθείτε σε πολύ βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Γιατί όλη αυτή η δουλειά με το εξάμεινο, ξέρετε, ε, και, και θα ήθελα να ρωτήσω και τι είδους ε, συστάσεις θέλετε να μας υποβάλλετε για τον ε, διάλογο αυτόν που θα αναπτύσσετε μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής και ιδιαίτερα όσον αφορά την αποδοχή και την αποδοτικότητα των μέτρων και είμαστε στο πλαίσιο του BRD, του ενιαίου ψηφίσματος, ε, τα κοινά ταμεία, ε, πιστοτικές δυνατότητες από κοινό ταμείο για την Ευρωζώνη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν έχετε κάποιες συστάσεις, προτάσεις και για το θέμα αυτό, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον από εσάς να ακούσουμε μια γνώμη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. και τον Ζωπολ και την Ελίζα ευχαριστώ πολύ για τα γενικά σας λόγια. Βεβαίως, στο θέμα του εξαμήνου, του οικονομικού εξαμήνου έχουμε πολλά να πούμε. Είναι πιστεύω μια καλή διαδικασία με περισσότερη πειθαρχία, πιο έγκαιρη εκκίνηση από την μελέτη ανάπτυξη στο οικονομικό πρόγραμμα που ετοιμάζουμε εμείς τώρα. Και βέβαια με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος. Έχουμε σε σχέση με αυτό ε, κάποιες δυσκολίες και δεν ξέρω άλλες χώρες πώς ε, τα πήγαν στην υπόθεση αυτή, αλλά το εξήγησα και στο Συμβούλιο ότι οι προϋπολογισμοί συνήθως είναι πιο κλειστοί, δεν είναι τόσο διαφανείς ως προς τις προβλέψεις για ε, φορολογικά έσοδα. Ωραία. Εμείς λοιπόν τώρα στη Μάλτα το κάναμε, κρίναμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού, δημοσιονομικού προγραμματισμού και προβλέπουμε ένα συγκεκριμένο ποσό από ειδικού φόρους. Ε, Αμέσως λοιπόν βγήκανε τα άρθρα για τους προβλεπόμενους φόρους ε, σε τσιγάρα, αλκοολούχα κτλ. Και μέσα σε μερικές εβδομάδες αδέσαν τα ράφια των καταστημάτων από αυτή την κερδοσκοπία που προέκυψε μόνο και μόνο από την ανακοίνωση των προθέσεων. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση δεν οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα τη Μάλτα. Κατά τα άλλα, και τα σχεδιαγράμματα που έπρεπε να ακολουθήσουμε ήταν χρήσιμα. Μαθαίνουμε πάντως. Ήταν μια πρώτη εμπειρία αυτή. η Υπουργοί των Οικονομικών σε συνεργασία, συντονισμό των προϋπολογισμών και βέβαια με όλα αυτά τα παραθυράκια που εξετάζαμε και συμπληρώναμε ανάλογα με τον κίνδυνο. Μαθαίνουμε λοιπόν και η αίσθηση που έχω, και ήταν κύρια που είχα εξ αρχή με τον Όλυ Ρεν, ε, αυτό του είχα επισημάνει, ναι αφήστε με να το κάνω μεν, να το κάνω, να το αναλάβω, αλλά και σε μια ε, αίσθηση αυτοσεβασμού. Μην ε, φαίνεται, όπως και με την Ιταλία και με τη Γαλλία, μην ακούγεται ότι α, το έκανε η κυβέρνηση γιατί το επέβαλε η Επιτροπή, γιατί πολιτικά ξέρετε αυτό δεν έχει καλά αποτελέσματα. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει εν τέλει, ότι υποσχεθούμε να προσφέρουμε και σαν αποτέλεσμα. Αυτά νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Επίσης ο συντονισμό ε, των ε, προπολογισμών δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Η Ιρλανδία φέρει πήρε ανακοίνωσε προπολογισμό. πέρασε στη διαδικασία την κοινοβουλευτική αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Εμείς Έχουμε κάποια θέματα τα οποία χρειάστηκε την τελευταία στιγμή να εγκρίνουμε παρότι είχαμε συζητήσει με την Επιτροπή. λέγαμε δράση όταν μας είπαν ότι αυτό δεν αρκούσε. Αυτό που είχαμε προβλέψει και κατά κάποιο ποσοστό ήταν ανεπαρκές, ήταν ελλειπές και άρα μέσα σε, σε μια-δύο εβδομάδες κάναμε τις προσαρμογές. Και μάλιστα υπήρχαν οι σχετικές αναφορές στον τύπο ότι η Μάλτα όχι για την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, αλλά για τον προπολογισμό του 2014 έκανε τις προσαρμογές κτλ. Για την Τραπεζική Ένωση είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους, διότι αναφέρεται στο μέλλον αυτό. Και θα θέλαμε βέβαια περισσότερη ευελιξία. Η ευελιξία όμως βοηθάει τις πιο μικρές χώρες ή τελικά τις πιο μεγάλες μόνο να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες. Πολύ δύσκολα ζητήματα. Έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και σκοπεύουμε να το διατηρήσουμε, να το διαφυλάξουμε. Ε, γιατί όταν μιλούμε για σωστούς, ε, σωστές αναλογίες, ε, κεφαλαιοχικές απαιτήσει. προφανώς κανείς δεν θέλει να γίνει σεισμός, αλλά σεισμοί συμβαίνουν. Και η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν διαστάσεων εγκέλαδου για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ε, για τον ένα λόγο ή τον άλλον, μπόρεσαν οι τράπεζε στην ε, Μάλτα να ε, σταθούν στα πόδια τους, να μην επηρεαστούν, να μην χρειαστούν διάσωση. Και βεβαίως πολύ καλό είναι που δεν, συνέβη, που δεν αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε για το μέλλον και μόνο σε δείκτε μπορούμε να στηριχθούμε. Κάναμε τους υπολογισμού μα και είδαμε ότι οι τράπεζε μα είχαν επάρκεια να ικανοποιήσουν τι απαιτήσει. Συμφωνήσαμε λοιπόν μαζί τους. Το θέμα βεβαίως του ενίου ψηφίσματος δημιουργεί πιο πολλά προβλήματα με την Ευρωζώνη και την ομάδα της Ευρωζώνης και τους εκτός του ευρώ. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τη μια μέρα συνεδριάζουμε ως Ευρωζώνη, ε, Eurogroup, παίρνουμε τι αποφάσεις μας σε μια μεγάλη οικογένεια κτλ. Και μετά πάμε την άλλη μέρα σε μια μεγαλύτερη ομάδα, όπου η μεγαλύτερη ομάδα δεν ξέρει τι έχει αποφασιστεί την πρώτη μέρα. Γιατί δεν είναι παρόντες. Και δεν έχουν και το ESM ως ε, ε, δυσφαλιστική δικλίδα. Όλα αυτά προξενούν τριβές. Δηλαδή δεν λαμβάνονται αποφάσει από μία μόνο ομάδα που θα συμφωνήσει τα θέματα αυτά, αλλά από δύο χωριστέ. Κατά άλλα συμφωνούμε με την Τραπεζική Ένωση, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει, η εποπτική αρχή και για συστημικούς κινδύνους, όπω πολύ καλά γνωρίζουμε, χρειάζεται ε, ένα δίκτυο και κάποια κεντρική παρακολούθηση και υποπτία. Και άρα, ναι, δεν θέλουμε να παρελκύσουμε τις εξελίξεις, δεν θέλουμε να προξενήσουμε καθυστερήσεις. Είναι μια εξέλιξη, ένα μέτρο το οποίο περιμένουν και οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και πρέπει να συμφωνήσουμε ή μη τι άλλο στο σχέδιο, το, το φύλλο πορείας, όπως θέλετε να πείτε το. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε προσχήματα για να καθυστερήσει αυτή η υπόθεση. Δεν πρέπει να καθυστερήσει. Κυρία Μπόλς. Ε, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Θα ρωτήσω μια συμπληρωματική ερώτηση και στο θέμα ιδιαίτερα της νομοθεσίας που κρίνεται σαν, ε, σε επίπεδο ένωσης. Είπατε ότι συνεδριάζετε σε, στο Eurogroup, παίρνετε τις αποφάσεις και αυτό το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να πει αυτή την ομάδα αν εγώ δεν ήμουν στο ευρώ, τι συνέπειες θα είχε και σε ποιο βαθμό μπορούν οι υπόλοιποι που είναι εκτός αυτής της αίθουσας τώρα να αποδεχθούν τις αποφάσεις για τη διαδικασία για τις τράπεζες. Έχουμε να κάνουμε μια από τις αρχές ε, του FSP και νομίζω και ακόμα και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συζητάμε. Μπορεί βεβαίω αυτοί που δεν ανήκουν στο Eurogroup να είναι ο μεγάλο απόν, του οποίου βαρύνει η παρουσία, η απουσία μάλλον από την αίθουσα, αλλά πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στι αποφάσει που λάβετε στο Eurogroup. Δεν είπα ότι δεν το εξετάζουμε, αλλά είπα ότι είναι μια επιπλέον επιπλοκή και θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη, γιατί είναι κάτι που είναι σταθερό. Και κάθε φορά που μια χώρα, Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή, η Πολωνία έχει αντίρρηση, έχει αντιδράσεις, το σκεφτόμαστε. Και την τελευταία φορά στην Ιρλανδική Προεδρία είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Περάσαμε μια ολόκληρη νύχτα, δεν ξέρω τι ώρα τελειώσαμε, στις 8 το πρωί, αλλά εξακολουθούσαν η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο να υποβάλλουν ενστάσεις. Τελικά υπέκυψαν και έκλεισε η συμφωνία, αλλά πρόκειται κάτι που ισχύει, είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και να μην την αγνοούμε. Ευχαριστώ, Σβέν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω καταρχήν, όχι μόνο στο Twitter, αλλά και αυτοπροσώπως. Μετά τους συντονιστές ε, είχαμε μια πολύ διασκεδαστική ελληλογραφία και είχε πλάκα γιατί ε, η γραμματεία μου είπε δεν, ήταν δεν είναι εύκολο να βρούμε εκείνη η ημερομηνία αλλά εγώ τους σου στείλα μέσα ένα tweet και τα καταφέραμε. Θα πρέπει να πείσουμε τη γραμματεία να χρησιμοποιεί το Twitter γιατί είδατε τι εύκολα βρήκαμε τελικά μια κοινή ημερομηνία. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ακούσαμε την ενημέρωση για τον προϋπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περίφημοι πίνακες αντιστοιχίες ή συγκριτικές στήλε που δημιουργήθηκαν γιατί το Κοινοβούλιο επέμεινε να έχουμε πιο συγκρίσιμα μέτρα και βλέπετε ότι η χειρότερη χώρα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση των ειδικών στάσεων αναχώρα είναι η Γερμανία συμμορφωση των ειδικων στασεων αγαναχωρα ειναι η Μάλτα έχει τη βάση ουσιαστικά στη βαθμολογία. Μέτρια πρόοδο δηλαδή. Ε, τώρα, έχουμε περιορισμένη δράση στα συνταξιδοτικά συστήματα. Ενημέρωση σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση στο δομέα της υγείας, που δεν είναι ικανοποιητική, ανεπαρκής, αυτό λέει η Κομισιόν. Και επίση ε, υπάρχουν κίνδυνοι έγκριση και εφαρμογή σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση της αποτελεσματικότητας ε, στη δημόσια διοίκηση. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτά τα εδάφια. Και έχω και μια άλλη συγκεκριμένη ερώτηση που συχνά απασχολεί και τον τύπο. Βέβαια είναι προφανές ότι έχετε δημοσιονομικά προβλήματα και οι προβλέψεις του φθινοπόρου δείχνουν ότι η διαθροτική ισορροπία για το 2013 και 2014 διατρέχει κίνδυνο. με 650.000 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει τη και Θαγένεια. Χωρίς καν να χρειάζεται να ζει ή να επενδύει στη Μάλτα. Ουσιαστικά πουλάτε πρόσβαση σε μία χώρα που είναι στην Ευρωζώνη. Η Ιθαγένεια χώρες στην ευρωζωνη η χώρα της ευρωζωνης και το κάνετε μόνο για τα χρήματα. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις γιατί ε, το θέμα απασχόλησε και τη Γερμανία. Είναι ασυνήθιστο να μπορεί κανεί να αγοράζει την ηθαγένεια μια χώρα χωρί καν να διαμένει στη χώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δίνεται ηθαγένεια σε αλλοδαπού, αλλά τουλάχιστον να έχουν πραγματικού δεσμού με τη χώρα. Γιατί λοιπόν το κάνετε. Γιατί η διόρθωση της τρύπας του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να γίνεται με την ε, εκποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση, Βέν, γιατί αυτή είναι και πιο σημαντική. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό δεν είχε καμία σχέση με το έλλειμμα ή με τα οικονομικά μας. Ο γραμματέας μου είναι εδώ και το συζητήσαμε και σχεδόν το αποκλείσαμε γιατί είπαμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει μόνος του να στέκεται στα πόδια του. Και τελικά ε, είπαμε 15 εκατομμύρια. Η Κομισιόν είπε να το μειώσουμε στα 8 εκατομμύρια σε ένα προπολογισμό 3,5 δισεκατομμύρια. Βέβαια, 3,5 δισεκατομμύρια για μεγάλε χώρε δεν είναι τίποτα, αλλά μιλάμε για την Μάλτα. Οπότε 8 με 15 εκατομμύρια είναι ένα δείγμα. Είναι πολύ μικρό τμήμα ο προπολογισμό στέκεται και χωρί αυτό. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτό το μέτρο δεν συνδέεται με το έλλειμμα ή με τη διόρθωση, την κάλυψη της, του προπολογισμού. Και αναφέρεται αυτό το 3,4-3,5 που στηρίζεται στην, στο τεκμήριο ότι θα ληφθούν φόροι από την κατανάλωση. Αλλά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Το θέμα είναι ότι τα επενδυτικά μας προγράμματα δεν είχαν σχέση με το θέμα αυτό. Οι επενδύσεις όμως μας ενδιαφέρουν και χαίρομαι που το αναγνωρίζω και δημοσίως. Το θέμα ξεκίνησε με την πρόταση για την ε, ίδρυση μιας αναπτυξιακής τράπεζας στη Μάλτα. Ναι, το έλλειμμα φυσικά μετράει, βαρύνει. Και η κυβέρνηση με την ε, δημοσιονομική διακυβέρνηση και με την περικοπή του ελλείμματος στο κάτω από τα 3% έχει δεμένα χέρια ουσιαστικά. χρειαζόμαστε κάποιον άλλο μηχανισμό για να διαχειριστούμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Έχουμε πολλές τράπεζες εμπορικές, αλλά θέλαμε ένα μηχανισμό για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαβουλεύθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έγινε μια πρόταση, αλλά αυτό είναι ένα, μια λύση, καμία σχέση με την IIB. Άλλη λύση ήταν ότι και εμείς όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, να έχουμε ένα σύστημα ώστε ένα καθεστώς όπου όσοι επενδύουν στη Μάλτα να μπορούν να να μπορεί να αναγνωρίζεται αυτή τους η προσπάθεια. Αλλά ήταν δύο τελείως ξεχωριστά πράγματα. Τώρα, με δημόσιο διαγωνισμό ζητήσαμε συμβουλές από, μια από ένα ανεξάρτητο γραφείο που είχε διεθνώς αναγνωρισμένη πείρα και αυτή η ομάδα έκανε το μάρκετινγκ και πρότρεξε ουσιαστικά σε σχέση με αυτό που έπρεπε να κάνει η τράπεζα ή το επενδυτικό ταμείο. Και γι' αυτό έφτασε αυτή η είδηση. Και εγώ το ακούγα αυτός ο Ευρωβουλευτής ότι οι Μαλτέζοι πουλάνε ένα διαβατήριο για λεφτά. Φυσικά ακούγεται ανάρμοστο. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτή η εντύπωση δόθηκε, ήταν ατυχής και διορθώθηκε τελικά. Καταρχήν δεν υπάρχουν νομικά σημειώματα με λεπτομέρειε δεν δημοσιεύτηκε τίποτα τέτοιο. Ο Πρωθυπουργό έχει συνάντηση με τον αρχηγό της αντιπολίτευση και συνεχίζονται οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα και η ομοφωνία που προτάθηκε, η εμπιστευτικότητα, η εμπιστευτικότητα μάλλον, το απόρριτο που ζητήθηκε από τους ε, ενδιαφερόμενους ε, απορρίφθηκε και Κάνουμε πολλές μεταρρυθμίσεις ε, σε πολύ λίγο χρόνο και συμφωνώ μαζί σας ότι για το θέμα αυτό θα, δεν θα έπρεπε να είχαμε δείξει τόση βιασύνη. Καταρχήν, ακόμη και η Μάλτα, μια μικρή χώρα, δίνει χίλιες ε, ηθαγένειες το χρόνο, κυρίως ε, λόγω γάμου. Δεν εξετάζουμε εξονυχιστικά αν κάποιος παντρεύεται από αγάπη ή απλώς για το συμφέρον του για να βρει δουλειά. Δεν δείχνουμε την ε, δέουσα επιμέλεια και μετά από τρία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε διαζύγιο που σημαίνει ότι κάποιος παντρεύτηκε μόνο και μόνο για να λάβει την υποκότητα. Πάντως ε, μας ενδιαφέρουν οι καλόπιστοι επενδυτές και 10 ή 15 ουσιαστικά όπως σας είπα εκατομμύρια. Δια 6, κάτι. 20, θα, 20 ουσιαστικά διαβατήρια σε σχέση με τα χίλια που δίνουμε κάθε χρόνο. Δεν θα έχουμε μαζική ε, συρροή Μαλτέζων υπηκών στην Ευρώπη με αυτά. Δεν ισχύει λοιπόν ότι όλοι οι Κινέζοι θα έρθουν στη Μάλτα, θα αγοράσουν ε, μαλτέζικο διαβατήριο και θα εισρεύσουν, ε, θα κατακλείσουν την Ευρώπη. Αλλά θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, θέλουμε περισσότερους δεσμούς, ε, όχι μόνο να γίνονται επενδύσεις, αλλά και να διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι στην Μάλτα και να αγοράζουν και όλα ακίνητα. Και πιστεύουμε ότι η Μάλτα μπορεί να είναι ελκυστικός τρόπος ο τόπος ε, διαμονής. Αλλά ελπίζουμε να μην είναι και μόνο για φορολογικούς λόγους, για ποδοσφαιριστές ή άλλους υψηλούς εισοδηματίες, για παράδειγμα. Θέλουμε τα χρήματα να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις και το Ταμείο των επενδυτικό αυτό το, το καθήκον θα έχει. Ήταν λάθος, επαναλαμβάνω, που δόθηκε αυτή η εντύπωση και πραγματικά δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις. Τώρα για το πρώτο τμήμα της ερώτησης, για την υγεία, τις συντάξεις και την αποτελεσματικότητα. Και αυτό το θέμα είναι δυναμικό και ένα μήνα μετά τις ε, εκλογές ξεκινήσαμε μία αξιολόγηση της κατάστασης ε, στα νοσοκομεία, στον τομέα της υγείας. Είδαμε πολλές αδυναμίες, σενάρια τρόμου, σε πολλές χώρες βέβαια παρατηρούμε τέτοια σενάρια τρόμου δεν είχαμε κεντρικό φορέα αποθήκευσης, πολλά προβλήματα σε νοσοκομεία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε έκθεση την περασμένη εβδομάδα και θα το συζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Το ίδιο και με την έκθεση για την μεταρρύθμιση τομέα της δικαιοσύνης. Όλα αυτά βρίσκονται εν εξελίξη. Δεν είναι απλώς υποσχέσεις, αλλά είναι διαδικασίες που συνεχίζονται. Και περιμένω και το δικό σας σχολιασμό. Και τον Απρίλιο ε, για, τις, ε, για τις Όλε αυτέ όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν υποσχέσεις. Τώρα έχουν εφαρμοστεί, έχουμε υποβάλει τον προϋπολογισμό. Και του χρόνου ελπίζω να έρθω και να σας ενημερώσω για το βαθμό στον οποίο ήταν αποτελεσματικές όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στο Κατζιάι. Έχουμε τον Πίτερ Σκίνερ και μετά τον Λίαμ. Ωραία. Λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι για να προλάβουμε. Πίτερ, ευχαριστώ πολύ. Έντουαρντ, ε, χαίρομαι που σε βλέπω όπως πάντα. Συγχαρητήρια νομίζω για τον ισορροπημένο προϋπολογισμό σας. Όποιος διαβάζει σχετικά ξέρει ότι ε, στην Μάλτα έγινε ε, έτσι, η διαδικασία επειδή στηρίχθηκε και τις δύο πλευρές του Κοινοβουλίου. Εδώ γίνεται λόγος και για κοινωνική οικονομία. Η μείωση του φόρου εισοδήματος ήταν σημαντική και ενδιαφέρουσα ε, ενέργεια, γιατί σε καιρούς λιτότητα συνήθως οι κυβερνήσεις κάνουν το αντίθετο. Είναι αυτό το τμήμα της, των προγραμμάτων ε, εγγύηση για την νεότητα ε, ή για την πρόθεση της δημιουργίας θέσης απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης. Και το δεύτερο στοιχείο που με ενδιαφέρει πολύ και υποψιάζουν πως όλοι πρέπει να κάνουμε την ίδια πορεία, ορισμένοι δεν αντιστέκονται ακόμα. Εσύ Ποιο θεωρείς ότι είναι τα πλονεκτήματα του τρίτου πυλώνα στην κατεύθυνση που εσείς διαλέξατε και τι κάλυψη νομίζω πως θα έχετε στην Μάλτα. Ευχαριστώ Πίτερ. Όσον αφορά την περικοπή του φόρου, θα είναι ουδέτερη. Δεν είναι μια περικοπή όπου θα, χαθεί, θα χαθούν έσοδα. Πρόκειται για μετακίνηση από άμεση φορολογία σε έμεση. Χοντρικά η Μάλτα έχει έσοδα από έμεση και άμεση φορολογία. Αλλά επίσης πρέπει κανείς να βλέπει και την κατανομή των εισοδημάτων και γνωρίζουμε ότι όπως σε πολλές χώρες, πολλές χώρες η κατανομή των εισοδημάτων επιδεινώνεται. Στην Μάλτα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το ποσοστό της στόχιας στη Μάλτα είναι ένα από τα χαμηλότερα, αλλά επιδεινώνεται. Ε, και αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Μόλις αυτή τη εβδομάδα συνάντησα τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και τώρα κοιτάζουμε ήδη τον προπολογισμό του 2015 ε, να δούμε στο χαμηλότερο μέρος, δηλαδή παιδιά, φτώχεια, όλα αυτά πώς θα εξετάσουμε και τώρα προσπαθούμε ήδη να δούμε πώς θα το αντισταθμίσουμε. Για τις συντάξεις, η Μάλτα είναι μοναδική. Ε, με την έννοια όπως εξήγησα, η δικιά μας συμμετοχή είναι τόσο μικρή, τόσο χαμηλή, υπάρχουν τόσο πολλά περισσότερα από το βάρος δηλαδή της σύνταξης το φέρουν λιγότεροι άνθρωποι. Οι περισσότερες χώρες έχουν το ίμιση του πληθυσμού τους να εργάζεται. Εμείς είμαστε 40.000 ε, μείων. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε εκεί, η κατάσταση λοιπόν θα βελτιωθεί, τουλάχιστον αυτό είναι ένα ένας τρόπος να δούμε τα πράγματα. Έπειτα το ίδιο το, το, το χρέος μπορεί να θεωρηθεί ως παθητικό όπως και οι συντάξει. Το να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το χρέος εκεί όπου θέλουμε να το σταθεροποιήσουμε μέχρι του χρόνου και αν μετά αρχίσει να μειώνεται θα σημάνει και ελάφρυνση του, ε, του, του, βάρους για τις μελλοντικέ γενναίες. Ωστόσο, εάν έχουμε ένα κοινό, κοινή ομάδα εργασία μεταξύ του δικού μου Υπουργείου και του Υπουργείου Κοινωνική Πρόνοια και κάνουμε τέτοιε προβολέ και υπολογισμού, ότι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Γιατί, όπω εξήγησα, κανεί δεν θέλει να πληρώσει τώρα για το μέλλον. Αλλά όταν του λε, θέλει τα παιδιά σου ή τα εγγόνια σου να είναι φτωχά όταν θα πάρουν τη σύνταξή του, τότε η απάντηση είναι όχι. Και άρα αυτό του οδηγεί να κάνουν αυτό που αντιστέκονται να κάνουν ε, τους αρέσει είτε όχι. <laughs> Οπότε γίνομαι όλο πιο πολιτικός. Προσπαθώ να καλύτερα να πουλήσω τα δύσκολα πολιτικά μέτρα. Ε, μάλλον είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση που κάνει κανείς εδώ στην ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ, Σαρώνα. Συγχαρητήρια. Για όσα καταφέρνεις, Εντουάρ. Είχα την τιμή να αναλάβω το πακέτο των προτάσεων για τις στατιστικές που είχες εσύ επομιστεί. Και έχω ένα προβληματάκι, μια δυσκολία με την Κομισιό. Που κατόπιν τριμερούς διαλόγου που είχαμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο παρακολεί τις εργασίες μας και ενώ είχαμε ψηφίσει σε πρώτη ανάγνωστο κείμενο και υιοθετήσαμε πιστά όλες τις προτάσεις της δικές σου. Μείναμε πραγματικά πολύ πιστοί στις θέσεις σου, προτάσεις σου. Και βλέπω ότι είχες ε, με πολύ φιλόδοξο τρόπο εργαστεί στο θέμα αυτό. Η δουλειά σου ουσιαστικά αναγνωρίζεται δηλαδή χάρη σε αυτή την ε, ψηφοφορία. Βλέπω λοιπόν ότι για την εντολή που θα πρέπει να ανατεθεί στην Προεδρία του Συμβουλίου εν ώψη του προσεχού τριμερού διαλόγου, γιατί βέβαια πρέπει να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει τριμερή διάλογο, έχουμε μια σχετική μειοψηφία, μειονοψηφία, στην οποία δυστυχώ συγκαταλέγεται η Μάλτα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Ήξερα ότι είναι ένα θέμα το οποίο, ε, για το οποίο εσύ με ιδιαίτερα. Α, με πιάσατε. Ναι, και εγώ το ρώτησα. Και είπα αυτή είναι η θέση της Μάλτας. Ε, τώρα όμως που έχω τα ενία του φακέλου αυτού από πλευρά της κυβέρνησης θα το κοιτάξω πολύ προσεκτικά, ασφαλώς. Θα ήταν κρίμα. Γιατί οι στατιστικές είναι όπως τα πόδια ενός γίγαντα. Κάναμε τόση πολύ και χρήσιμη δουλειά με την... Ε, ε με το six pack, με το two pack, με όλα τα μέτρα. Και αν είναι πύληνα τα πόδια του γίγαντα, ξέρετε πολύ καλά ότι θα καταρρεύσει. Ε, αυτά είναι τα πόδια του γίγαντα, οι στατιστικές, και πρέπει να είναι γερά τα πόδια αυτά. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γιατί οι προβλήματα, οι αναθεωρήσεις, αέπι, λάθη, πάντα οδηγούν σε χειρότερες δυσκολίε. Και χθε ήμουνα σε μια παρουσίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας ε, για το δυναμικό απόδοτο παραγωγικότητα, το οποίο εμείς προβλέπουμε να αυξάνεται, ενώ η Επιτροπή μας λέει θα μειωθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ενώ έχουμε αύξηση τη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, έχουμε μέτρα υποστήριξη τη παραγωγική διαδικασία, δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε πώ η Επιτροπή ερμηνεύει διαφορετικά τα, ίδια στοιχεία. Η ανεξαρτησία πάντω των υπηρεσιών και τη Eurostat ασφαλώ έχει τεράστια σημασία. και μόνο έτσι μπορούν να κερδίσουν τον σεβασμό. Αυτό ήταν, αυτή ήταν μια δοκιμασία από την οποία χρειάστηκε να περάσω και εγώ στην πατρίδα μου. Γιατί διαγνώστηκε ένα πρόβλημα, ένα λάθος και χρειάστηκε και να αναλάβω την πρωτοβουλία να στήσω διερεύνηση ως υπουργό, αλλά και να κρατήσω αποστάσεις. Και έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσεις κτλ. Βεβαίω, θα κοιτάξω τι μένει να γίνει, θα το υποστηρίξω, θα μιλήσω και με τη γύρω όταν χρειάζεται και με το Συμβούλιο. όπου ελπίζουμε ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως αυτό να κερδίσει τη συμφωνία των μελών του Συμβουλίου. Θα, τα αφήσω, θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Ναι, άρα τώρα έχουμε και τον δικό μας άνθρωπο στο Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Δεν είναι και η πρώτη φορά βέβαια που ενημερωνόμαστε πως τα κράτη-μέλη ε, παρεμποδίζουν πράγματα τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο για τις στατιστικές και για το 2010 είχαμε το ίδιο στις προβλέψεις του 2010, αλλά καταφέραμε τελικά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίε. Ξέρουμε τι πάει να κάνει το Συμβούλιο, αλλά θα μείνουμε δυνατοί και ενωμένοι. Ευχαριστώ πολύ Σάρων και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον φίλο. Με χαρά σας βλέπω εδώ, ως και γείτονα εδώ και συνάδελφος που έχουμε συζητήσει τόσες φορές μαζί. Σας καλωσορίζω για την καινοτόμο λύση που βρήκατε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ξέρετε και ποιο είναι το ιστορικό μας και το έχουμε καταφέρει για το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως ε, και από την εμπειρία σας ως Ευρωβουλευτή, αλλά και τώρα από τη θέση σας ως Υπουργού, θα ήθελα να ρωτήσω τι βλέπετε να μπορεί να αλλάξει ή να πρέπει να αλλάξει για τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ Βρυξελών και κρατών μελών. Και ποιο θέμα θα ήταν το πιο κρίσιμο, ώστε να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή και οι συζητήσεις πιο ειλικρινέ ίσω προς την ε, αλληλεγγύη, γιατί εμείς, ξέρετε, στου σοσιαλιστές δημοκράτες ε, συζητούμε τα θέματα αυτά πολύ συχνά. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι περιοριζόμαστε μόνο σε συζητήσεις. Θα μπορούσα να έχω κάποια απάντηση. Θα εστιαστώ στη μία λέξη που χρησιμοποίησε στην αλληλεγγύη. Γιατί λαός των χωρών σαν τη Μάλτα μπερδεύεται. Και όταν λένε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε άλλες χώρες μέσω του μηχανισμού σταθερότητας, χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης και να βοηθήσουμε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα ή όποια το χρειάζεται, συμμετέχουμε ε, αυθόρμητα και μάλιστα με συμφωνία κυβέρνηση και αντιπολίτευση εγκρίνουμε τις σχετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο. Και μάλιστα η Μάλτα δίνει 3,3% του ΑΕΠ σε αυτά. Καταναλογία πολύ περισσότερα από άλλες χώρες. Έχουμε δώσει πάνω από 3,3% του ΑΕΠ μας αυτό το προσωρινό και τα μόνιμα ταμεία και τους μηχανισμούς. Και μάλιστα όταν, αυτό σημαίνει επειδή είμαστε σε μεγαλύτερη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνήθω υπάρχει ένα κατώτατο όριο και ένα ανώτατο όριο. Μερικέ φορέ αυτό ο σχετισμό μα εξυπηρετεί, όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχουμε καλή εκπροσώπηση. Αλλά έχουμε και την αρνητική πλευρά, που είναι η συμμετοχή, η συνεισφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, με τον επιμερισμό του βάρους, εκεί αισθανόμαστε ξεχασμένοι, απομονωμένοι γιατί έρχονται οι μετανάστες σε εμά γιατί ε, είτε αναζητούν άσυλο, είτε προσπαθούν να, να ξεφύγουν από κινδύνους που διατρέχουν στη χώρα τους, ε, διακινδυνεύουν τη ζωή τους, ε, το γνωρίζουμε. Αλλά εκεί έχουμε μείνει τελείως απομονωμένοι, όχι μόνο η Μάλτα. Μένονται, μένουν απομονωμένοι και αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν πολλές φορές τη ζωή τους στη θάλασσα. Γιατί μερικές φορές ερμηνεύεται διαφορετικά η αλληλεγγύη. Και όλες αυτές οι διαφορές ε, δημιουργούν μια αδιαφορία του πολίτη για τις εκλογές. Βέβαια στη Μάλτα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε εκλογές, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και στις άλλες χώρες. Η Μάλτα δεν διαφέρει από τις άλλες χώρες. Υπάρχει υπάρχει μερικές φορές ένα γεφύρωτο κενό, μια γεφύρωτη απόσταση του κόσμου από την πολιτική. Και δεδομένη τη κρίση, ίσω θα μπορούσαμε να βρούμε αυτή την ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε την ελληνική και για να ενισχύσουμε την αλληλοβοήθεια, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Εν κατακλείδη, πάντως, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε θετικοί. Έχουμε πολλά φιλόδοξα σχέδια μερικές φορές ίσως ε, δεν υπάρχει, καλή κατανο... αλληλοκατανόηση, αλλά δεν υπάρχει μια λύση που εξυπηρετεί όλους. Δεν λέω ότι οι μικρές χώρες έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή θα πρέπει να τύχουν ειδική μεταχείριση, αλλά υπάρχουν διαφορές. Χθες διάβασα στην αφημερίδα ότι είναι διαφορετικά καλωδιωμένος ε, ο γυναικείος εγκέφαλος από τον ανδρικό εγκέφαλο. Είπα διαφορετική καλωδίωση και διασύνδεση των ευρώνων. Δεν λέω ποιο εγκέφαλο είναι καλύτερο των γυναικών ή των ανδρών. Το ίδιο ισχύει για τι χώρε λοιπόν. Δεν μπορούμε να τι βάλουμε όλε στο ίδιο καλούπι. Οπότε η προσπάθεια που αναμένεται από εμά με τι στατιστικέ, με, ε, με τα διάφορα θέματα, οι προσπάθειε που αναμένονται είναι τεράστιε. Και οι μικρέ χώρε, οι νησιά, είναι σε δυσμενή θέση. Αλλά είμαστε παρόλα αυτά και εμεί κράτο, κυρίαρχο κράτο και τη χάνουμε ίση μεταχείριση με τη Γερμανία. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε και εμεί στα πόδια μα και να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει. Ελπίζω πάντως να είμαστε πιο ευέλικτοι τελικά και ελαστικοί σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των χωρών. Ειδικά τώρα που είμαστε 28 Φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μελετήσει 28 προπολογισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να τσεκάρει όλα τα κουτάκια. Ε, λάθη γίνονται. Μόλις τώρα δημοσιεύθηκε μια έκθεση που αναγνωρίζει σφάλμα. Το 30 έγινε 300, το 40 έπρεπε να γίνει 400, έπρεπε να γίνουν διορθώσεις. Πάντω, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε σήμερα εδώ. Ε, βεβαίως, ε, κανονικά όλοι πρέπει να γίνουν ε, μέλη της ΕΚΟΝ πριν να γίνουν Υπουργοί Οικονομικών, γιατί έτσι παρουσιάζουν τα πράγματα με τρόπο που να αντιλαμβάνεται ο κόσμος και αντιλαμβάνεσαι καλύτερα ποια είναι τα θέματα ανάμεσα στα κράτη-μέλη με διαφορετικά μεγέθη. Και αυτό μας έδωσε και εμάς μια σαφή εικόνα για το τι διακυβεύεται από την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ.